Τα αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 32 υπέρ. Κατά αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο. Για την 32 της Επιτροπής Ανάπτυξης αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. So we come to compromise. Προχωρούμε. Συμβαστική 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 268 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 15 τώρα υπέρ κατά αποχές. Ξανά παρακαλώ υπέρ κατά είναι τα 15. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτς 3 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τι έγινε. Α, είχε καταπέσει, τώρα το σκοτώσαμε τελείω. Λοιπόν. 270... Α, όχι, έχουμε πρώτα το δεύτερο τμήμα και μετά τη 279. Λοιπόν, υπέρ του δεύτερου τμήματο τη μπάτση 3 κατά αποχέ εγκρίνεται. 279 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 280 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Μπάτζε 7 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα σε αιτιολογικέ σκέψει. Recycles. 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχέ. Τσεκ. Την 5 αιτιολογική σκέψη. Αρχίζει η ψηφοφορία και τελειώνει. Εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 14 παρακαλώ της κυρίας Πόστ. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. 29-27. Προχωρούμε στη 13 της ΔΕΒΕ. Υπέρ κατά αποχές. 80% των μελών δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Άρα χρειάζεται έλεγχος τώρα. ΔΕΒΕ 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 48-7. Εγκρίθηκε μάλλον. Προχωρούμε. Είναι τα τρία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα τέσσερα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθούν οι αιτιολογικέ αναφορέ. citations. Είναι τα ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, είναι τα δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμό 3 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ 4, 3 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Wow! Φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σχέδιο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. It's closed. Εγκρίθηκε. 42 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. We come to item number 9. Πάμε στο σημείο 9. Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εισηγητή τον Τζέφρι Βανόρντεν θέλετε να πείτε κάτι. Okay, but Ms. would like to say something, please. Η κυρία Νικίνη ήθελε να πει κάτι, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Λίγες παρατηρήσεις όσον αφορά την λίστα ψηφοφοριών του ΕΛΚΑ. Λόγω αλλαγών τη τελευταία στιγμή, ε, όσον αφορά τι απόψει ορισμένων πολιτικών ομάδων, η συμβιβαστική 5 παρακαλώ ψηφίστε όχι. Και στην τροπολογία 103 καταψηφίστε την. Αυτά. Ευχαριστώ. Okay, thank you. ευχαριστούμε. Άλλες παρατηρήσεις. Άλλες λίστες ψηφοφοριών πρέπει να αλλάξουν. Όχι. Ωραία. Τότε προτείνω να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Συμβεβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159 του κυρίου Μπούχνερ υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Πάμε στην 82. Σωστά του κυρίου Αντάκτουσον. Υπέρ, κατά, εποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ελέγχουμε την 85 του κ. Καστάλντο Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές. Θα έλεγα ότι εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 87. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά. 88 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 88 επίσης. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 90. Σαφχάουζερ υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 93-94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. 101 Σαφχάουζερ ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 να ελέγξουμε. κύριε Πρόεδρε. Δεν εγκρίθηκε η συμβαστική πέντε. Όχι. Ωραία, συγγνώμη. Εκατόν τρία πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 104, 102. Α, καταπίπτουν. Οπότε πάμε στην 102. Λαλόντρι και υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε την 150. Πέρα ψηφοφορία εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 156 αποσύρεται. 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 160 465 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 173, 75, 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι Πάμε στην 186 του κ. Σαφχάζερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 195 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 195 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 169. Όχι. «196 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204. Να ελέγξουμε τη 203 του κ. Μπούχνερ. The vote is closed. Oh. απορρίπτεται. 204 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205. Πάμε στην 13 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 13. 13. Ξεκινάει η ψηφοφορία. The vote is closed. Very clearly carried. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 21. Το open, Ξεκινάει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 24 πέτρελα ξεκινάει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 30-29 27 ε, υπέρ κατά εποχές να ελέγξουμε Πέτρα λεξανά, την 27 αρχή η ψηφοφορία. Ελέγξαμε την Πέτρελε θετικά λοιπόν, το θετικό το αποτέλεσμα. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε ξανά. 30 του κυρίου Αντάκτουσον. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφου. Είναι ο εδώ, όχι. Μην του πείτε τίποτα. 31. Κύριο Σοφχάουζερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεστική 1 υπέρ Συγγνώμη, την 34 την εγκρίναμε, οπότε πάμε στο κύριο επιτίδιο, 35 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κα... καταπίπτει 39, α όχι, 39 υπέρ, κατά αποχές, να ελέγξουμε την 39. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται κατά μία ψήφου. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 σαφχάζερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 51. Τρίτη φορά που ελέγχουμε τον κυριο πετρελα Πέτρελε. Πέρας ψηφοφορίας. 42-16. Με κάθε ψηφοφορία γίνεστε όλο και πιο δημοφιλής κύριε Πέτρελα 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 50 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 λάθος έκανε ο πρόεδρος 63 όχι 62 συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 σαφάζερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70-71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72. Υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε την 72 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται Σαφχάζερ ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 73 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 75 πέρας απορρίπτεται ήταν προφανές φαινόταν από εδώ 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά απορρίπτεται πάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου της γνωμοδότησης ξεκινάει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι 49 έναντι 5 υιοθετείτε πάμε τώρα στη σύναψη τη Συμφωνία Πλαισίου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη αφενό και τη Αυστραλία αφετέρου. Το συζητήσαμε χθε το απόγευμα. Ο εισηγητή, ο κ. Μιλανμόν, θέλει να πει κάτι. Όχι. Ωραία. Μπορούμε να προχωρήσουμε μέσω στην ψηφοφορία. Μία είναι Λοιπόν, αρχίζει τώρα για την Αυστραλία. Πρώτα θα ψηφίσουμε τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Όχι. Μα, τι ψηφίζουμε τώρα. Δύο συνάδελφοι δεν ψηφίζουν. Ένας τώρα. Όλοι ψηφίσατε. 55 υπέρ, 3 ε, αντίθετες ψήφοι. Και τώρα ε, πάμε στο σημείο 11 που είναι το συνοδευτικό ψήφισμα στην έγκριση σύναψη Τώρα θέλει να πει τίποτα ο κύριος Μιγιανμόν. Όχι. Προχωρούμε λοιπόν και πάλι στην ψηφοφορία. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ ότι είναι 25 επαληθεύουμε. αρχή ψηφοφορία. Απορρίπτεται. και 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35-36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. 38 είπε. κατά αποχές. Εγώ θα λέγω ότι έχει εγκριθεί τώρα αυτό. Το 38 εγκρίνεται, τι λέτε. Μάλιστα. 39 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ. Παληθεύουμε τη 48 του κυρίου Τάνοκ. Πέρασα. Απορρίπτεται. 49 του κύριου Επιτίδη επέ, κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Έλεγχος. Στη 17 είμαστε, του κυρίου Τάνοκ. Εγκρίνεται 37-22. 18 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 19 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να τσεκάρουμε τη 19, έτσι να έχουμε μια γεύση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και τελειώνει αμέσω. Δεν κρίθηκε. 20 είπε Πάλι όταν κατά αποχές εγκρίνεται. 21 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 22 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 23 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Τσάρλς πέντε νίκες σε σημείωση μόνος σου. Γι' αυτό δεν ήθελα να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Λοιπόν, citations 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο λοιπόν τώρα ηλεκτρονικά παρακαλώ η τελική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Πέρασε 54-2 συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Item number 12. 12 πρωτόκολλα τη Συμφωνία Εταιρική σχέση και συνεργασία για τη σύνευση Εταιρική σχέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών του Αφενό και τη δημοκρατία του, του Ουσμπεκιστάν αφετέρου ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση τη δημοκρατία τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσύγητης είναι ο κύριο Ράντο. Δεν ξέρω αν θέλετε να μα πείτε τίποτα περισσότερο. Απουσιάζει κιόλα, ωραία. Μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία ηλεκτρονική που αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 ψηφί, υπέρ με 3 δαρτά. Τελευταία ψηφοφορία του σημείο 13. Συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών τη αφενό και τη Δημοκρατία τη Κορέα αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση τη Δημοκρατία τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Τοκιά Σαΐφη είναι η συγγήτρια. Δεν θέλετε να μας πείτε τίποτα κρίμα. Ωραία, ας ψηφίσουμε λοιπόν αμέσως. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και τελειώνει. Ε, 57 υπέρ 3 ψήφοι κατά. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Τα ξεπετάξαμε. 10 λεπτά νωρίτερα. Αλλά έρχεται υπουργό. Έχουμε υπουργό εξωτερικών της Νορβηγίας. Καλό θα ήταν να παραμείνουν ορισμένοι από εσά τουλάχιστον για την ανταλλαγή απόψεων.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 Right, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι ακριβώς 10 η ώρα και με μεγάλη μου χαρά και τιμή, τιμή για όλους μας, ε, καλωσορίζουμε την κυρία Είναι Έριξεν Σέραϊντ, η Υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας. Την καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας Θυμάμαι ότι ο προκάτοχό σα ε, ήταν σε αυτή τη... είχε επισκεφθεί την επιτροπή μα. Και πάντα είναι ευχαρίστηση για μα να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπου τη νορβηγική κυβέρνηση που με του οποίου συνεργαζόμαστε σε τόσο πολλά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Δεν μπορώ να σα πω πολλά, δεν χρειάζεται για τη στενή μα ε, διμερή συνεργασία. Με καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχουμε τόσο στενέ σχέσει όσο με του Νορβηγού φίλου από τη συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας όσο και στη συνεργασία για περιφερειακά ζητήματα όπως την βιώσιμη ανάπτυξη, τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Εκεί πάντα η Νορβηγία συμφωνεί με τις δικές μας θέσεις. Για παράδειγμα όσον αφορά τη Ρωσία. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πολλά ζητήματα. Οι συνάδελφοι με βεβαίως ε, θα ακούσουν με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς η Νορβηγία σχεδιάζει να συνεχίσει τον δραστήριο ρόλο της στις πολιτικές Αρκτικής. Θυμάστε τι γεωπολιτικό βάρος, ολένα ένα αυξανόμενο, ε, παρουσιάζει η Αρκτική. Θα θέλαμε επίσης να μας πείτε κάτι όσον αφορά τη συνεργασία με την Νορβηγία στη γεωγραφική περιοχή ε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δυτικά Βαλκάνια, στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, ε, Χωρίς άλλη καθυστέρηση σας δίνω το λόγο. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ. Έχω ξαναέρθει στο παρελθόν, αλλά μόνο ως ακροάτρια για ανθρώπους που έκαναν ομιλίες εδώ. Ε, εγώ τότε ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μας ε, συχνά επισκεπτόμουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπως είπατε πολύ σωστά από το 1994 όταν ψηφίσαμε κατά του να γίνουμε μέλος ε, αποτελέσαμε τελικά μια από τις πλέον ολοκληρωμένες μη ευρωπαϊκές, μη ενωσιακές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε νομίζω η μόνη χώρα που ουσιαστικά απορρίψαμε δύο φορές το να γίνουμε μέλος, το 72 και το 94. Ποτέ όμως δεν απορρίψαμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν στενούς δεσμούς όσον αφορά τις αξίες και γεωγραφικούς. Η δική μας ασφάλεια και ευημερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δική σας. Οι ευρωπαϊκές δυσκολίες ε, είναι δυσκολίες και της Νορβηγίας και αντιστρόφους. Η νέα μας ε, κυβέρνηση, το συνόψε πολύ σωστά, είπε η εξωτερική πολιτική της Νορβηγίας ξεκινάει από την Ευρώπη. Και οι συναδελφοί μου και εγώ επισκεπτόμαστε συχνά τις Βρυξέλλες. Ενίοτε και πολλές φορές το μήνα. Ένα παράδειγμα της στενής μας συνεργασίας είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 20 υφυπουργού ε, και εκπροσώπους της ε, νορβηγικής κυβέρνησης εδώ σε συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, Συγγνωμένοι του Κοινοβουλίου μας. Θα σας πω δύο λόγια για το τι με έφερε εδώ σήμερα. Τις τελευταίες δεκαετίες η Νορβηγία και οι εταίροι μας της διεθνούς κοινότητας έχουμε επενδύσει σημαντικές διπλωματικές προσπάθειες και πόρους για την επίτευξη ε, βιώσιμης ανάπτυξης ε, στην ε, Μέση Ανατολή. Μετά από τη συμφωνία του 1993 του Όσλο, ακολούθησε η Επιτροπή την οποία εμείς προεδρεύουμε από το 1993. Βασιζόμαστε στη στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς ενδιαφερομένους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι λοιπόν να πιστεύω που μας φιλοξενεί στην ερνή συνεδρίαση η κυρία Μογκερίνη. Έχουμε λοιπόν και μια συνάντηση αργότερα σήμερα και σκοπός της συνάντησης είναι να συμφωνήσουμε επί κάποιων στρατηγικών μέτρων που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους παλαιστινιακούς θεσμούς και θα τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη, ειδικά στην Δυτική Γαζά, όπου, στη Δυτική όπου η κατάσταση είναι δραματική αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν γίνει άμεσες συνομιλίες εδώ και μια τετραετία. Αυτές οι συνομιλίες πρέπει να επανεκκινηθούν, αλλά πρέπει να θέσουμε και τα θεμέλια για να ξεκινήσουν τέτοιες συνομιλίες. Στην εκτέκτη συνάντηση της 31ης Ιανουαρίου εδώ στις Βρυξέλλες είχαμε την πρώτη συνάντηση ουσιαστικά μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων μετά από την δήλωση των ΗΠΑ ότι θα μετακινούσαν την πρεσβεία του στην Ιερουσαλήμ. Το επίπεδο συμμετοχής και η επικοδομητική, το επικοδομητικό περιβάλλον ε, του οργανισμού δείχνει δείχνει ότι πρόκειται για έναν σημαντικό μηχανισμό, έναν από του ελάχιστου μηχανισμού που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή, ώστε τα μέρη ε, και οι χορηγοί της ίδιας ε, της διεθνούς κοινότητας να κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι με στόχο τη διαπραγμάτευση ε, μιας λύσης με δύο κράτη. Σκοπός του οργανισμού είναι η επίτευξη προόδου επιτόπου, η πρόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και η ενίσχυση των Παλαιστινιακών θεσμών. Η AHLC είναι το μόνο διεθνές φόρουμ όπου συμμετέχουν ε, όλα τα μέρη και υπάρχει διάλογος και με τους ε, χορηγούς και με τη διεθνή κοινότητα. Αυτή την εβδομάδα η σύρεξη στη Συρία μπήκε στην 8ο έτος της και η φρικεστική κατάσταση στην Ανατολική Γούτα μας υπενθυμίζει σε όλους ότι ε, δεν έχει ακόμη τελειώσει αυτός ο πόλεμος, μακράν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας λοιπόν θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για μια βιώσιμη ανθρωπιστική εκεχηρία ε, κρίσιμη σημασία για να μπορέσει να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια, να εκενωθούν οι τραυματισμένοι και να προστατευτούν οι άμαχοι. Παρότι ιτήθηκε το ISIS ε, στρατιωτικά, εγώ ανησυχώ για την κλιμάκωση του τελευταίου μήνα. ειδικότερα στα βορειοδυτικά μέρη της Συρίας. Η διεθνή συμμετοχή στη σύραξη αυτή είναι ανησυχητική εξέλιξη. Η κατάσταση στο Αφρίν είναι δραματική. Μετά από την εισβολή της Τουρκίας τα αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα, αβέβαια. Όπως ξέρουμε όλοι, οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Συρία είναι γιγάντιες. 13,1 εκατομμύρια άνθρωποι χρήζουν ανθρωπιστική βοήθεια εντό τη Συρία, και 5,5 εκατομμύρια έχουν φύγει ως πρόσφυγε. Την τελευταία οκταετία η Νορβηγία έχει παράσχει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στη Συριακή κρίση και στη διάσκεψη του Λονδίνου του 2016 υποσχεθήκαμε και άλλα χρήματα για την επόμενη τετραετία σε ανθρωπιστική βοήθεια. Το 2018 λοιπόν θα παράσχουμε 225 εκατομμύρια ευρώ στη Συρία και στι γειτονικέ χώρες. Οι προτεραιότητε μας είναι η ανθρωπιστική αρρωγή και η παιδεία, ειδικότερα ε, για τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκε. Υποστηρίζουμε τις διαμεσολαβητικέ προσπάθειες των ΗΕ και στεκόμαστε στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα υποσχεθούμε συμβολή για την ανοικοδόμηση της Συρία μέχρι ότου θα έχουμε μία ε, διαδικασία ανοικοδόμησης ε, χωρίς αποκλεισμού. Αν πάμε τώρα στη Βορειοαφρική και στην περιοχή του Σαχέλ, έχουμε σημαντική παρουσία της Νορβηγία στην περιοχή. Συνεργαζόμαστε στενά με την Τινησία, με το Μάλι, με τον Ήγηρα και τον περασμένο μήνα ανοίξαμε την πρεσβεία μα στον Παμάκο. Η κατάσταση στο Μάλι και στην Λιβύη αποσταθεροποιεί την περιοχή στο σύνολό τη. Η ασφάλεια στη Βόρεια Αφρική και στην περιοχή του Σαχέλ, όπω γνωρίζουμε, είναι επίση σημαντική και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η αντιμετώπιση του βίου των διασυνοριακών εγκληματικών δικτύων τη ε, εμπορία ανθρώπων, όλα αυτά εξαρτώνται από τη σταθερότητα και τη συνεργασία. Η ειρήνη είναι κρίσιμη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τι επενδύσει του ιδιωτικού τομέα και για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, ε, σημαντικού παράγοντε ε, σε όλε αυτέ τι χώρε τη περιοχή. Θα υποστηρίξουμε την δύναμη των G5 ε, στο Σαχέλ για την οικοδόμηση δυνατοτήτων και για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε τη συμμετοχή μας στα πολυεθνικά ε, στρατιωτικά αεροσκάφη που ξεκίνησε η Νορβηγία και συμφωνούμε με την ηγεσία που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Οι κρίσεις ε, και οι σειράξεις στα πρόθυρα της Ευρώπης αυξάνουν την μετανάστευση προς την Ευρώπη. Εμείς ε, συμμετέχουμε στην απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεταναστευτικά θέματα πέραν της συνεργασίας Σέγγεν. Ε, μας συμφέρει και εμάς να βρούμε βιώσιμες λύσεις και με την κρίση των διεθνών υποχρεώσεων και των κανονισμών ε, έχουμε δεσμευτεί επίσης. Οπότε για μας αποτελεί όλο αυτό προτεραιότητα. Ε, συμφωνούμε με τη δημιουργία της Task Force για την προστασία των μεταναστών, για την επιστροφή ανθρώπων στι χώρε καταγωγή του και για την προστασία των ανθρώπων που χρήζουν διεθνού προστασία. Θα πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο που παρατηρούμε στη Λιβύη και ε, συμμετέχουμε και εμείς στο Trust Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να δώσει κατά προτεραιότητα βοήθεια στις πιο ευάλωτες ομάδες των προσφυγών. Ε, θα πρέπει να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τα πρότυπα του αυτό αποτελεί προπόθεση για τη δική μας χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε προτείνει να επαναγκαταστήσουμε 200.000 ε, και ε, μετανάστες το 2018, 300 από τη Λιβύη και αυτό σε στενή συνεργασία με το UNHCR. Ας πάμε τώρα στα Δυτικά Βαλκάνια. Η μεταναστευτική κρίση του 2015 σαφώς κατέδειξε αδυναμίες θεσμικές και άλλες στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Μας θύμισε όμως επίσης ότι είμαστε και αλληλένδετοι. Η σταθερότητα και η ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια είναι σημαντική για την Ευρώπη. Η αύξηση εθνικών εντάσεων και πολιτικών κρίσεων θα μπορούσε να διαδοθεί εύκολα στις γειτονικές χώρες. Η περιοχή απαιτεί ισχυρή ευρωπαϊκή δέσμευση και το στρατηγικό έγγραφο της Επιτροπής είναι επίκαιρο και η Νορβηγία συμφωνεί με τις προτεραιότητες του εγγράφου αυτού. Εκτιμώ ιδιαίτερα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι εκθέσεις πρόοδου κατά χώρα που προετοιμάζει η Επιτροπή θα διαβαστούν με μεγάλο ενδιαφέρον και εκτός της Επιτροπής αυτής. Και ο συνάδελφος, από το, ο συνάδελφος μου από το Κωσυφοπέδιο θα έρθει αργότερα σήμερα για να συζητήσετε τις σχέσεις ε, Κωσυφοπέδιου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη είναι σημαντική όχι μόνο για την ίδια την περιοχή αλλά και για τη μελλοντική ασφάλεια και ευημερία όλης της Ευρώπης. Η Νορβηγία υποστηρίζει ενεργά αυτή την ολοκλήρωση. Το 2018 λοιπόν θα διπλασιάσουμε την διμερή μας ε, βοήθεια στα Δυτικά Βαλκάνια σε περίπου 33 εκατομμύρια ευρώ το κράτος δικαίου, η ασφάλεια, η μετανάστευση, η ανάπτυξη είναι για μας τομείς προτεραιότητας. Επίσης υποστηρίζουμε τις επενδύσεις σε έργα υποδομής στα Δυτικά Βαλκάνια και στο σχετικό επενδυτικό πλαίσιο. Λόγω της σημαντικής μας δέσμευσης στα Δυτικά Βαλκάνια και της εστίασης σε προτεραιότητες επιπλέον των υπαρχουσών, ε, πιστεύουμε ότι όλο αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία στο μέλλον με την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα από τα Δυτικά Βαλκάνια στην Αρκτική. Στον... Είναι μεγάλο κομμάτι της χώρας μας. Σχεδόν το 10% του νορβηγικού πληθυσμού ζει εκεί. Εκεί ζει κόσμο, ξεκινάει επιχειρήσει, δημιουργεί επιχειρήσει, φτιάχνει οικογένειε και πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι η περιοχή τη Αρκτική είναι ένα παγωμένο μέρο, αλλά είναι μέρο που ζει κόσμο. Η Αρκτική. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Καθώ αλλάζει με ταχύ ρυθμού ο κόσμο, η Αρκτική αλλάζει όλο και περισσότερο. Και η κλιματική αλλαγή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Για να επιτευχθεί σωστή ισορροπία μεταξύ τη χρήση και τη συντήρηση των πόρων, απαιτείται επιστημονική συνεργασία. Αναγνωρίζουμε πόσο πολύτιμη είναι η συμβολή των Ευρωπαίων επιστημών στην καλύτερη κατανόηση τη Αρκτική. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ειρήνη, σταθερότητα και διεθνή συνεργασία και εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει έτσι. Τήρηση του διεθνού δικαίου, τήρηση του θαλάσσιου δικαίου είναι βασικοί παράγοντες και κανόνα στην περιοχή. Το Συμβουλίο της Αρκτικής, ε, η συνεργασία ε, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Θάλασσα Μπάρνς ε, αποτελούν διάβλους επικοινωνίας. Το Συμβουλίο της Αρκτικής είναι το βασικότερο διεθνέ όργανο για τη διαχείριση των ζητημάτων τη Αρκτική. Και εμεί το υποστηρίζουμε από πλευρά Νορβηγία και θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε με μόνιμη ε, παρουσία. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε παρουσία μόνιμου παρατηρητή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καταλάβει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχει δείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Η εργασία τη Επιτροπή σα ε, φαίνεται και στο σχετικό ψήφισμα που εθετήθηκε πέρυσι η δημιουργία του Φόρουμ Ενδιαφερομένων για την ακτική είναι ένα σημαντικό ε, ευπρόσδεκτο μέτρο. Στο βορρά έχουμε χερσαία και θαλάσσια σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Για μας η Ρωσία είναι ε, παγκόσμιος παράγων, αλλά είναι και γείτονά μας. Ως γείτονες λοιπόν επιδιώκουμε διμερή συνεργασία σε πρακτικά ζητήματα αμοιβαίων ενδιαφέροντος. Έχουμε πολλά διαφορετικά είδη συνεργασίας ο πιο σημαντικός τομέας συνεργασίας είναι η αλληλεία και η βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων μπακαλιάρου στην θάλασσα Μπάνζα, ε, ασφάλεια, διάσωση. Η στενή επαφή λοιπόν μεταξύ ανθρώπων είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής στο Βορρά. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε και υπερασπίζουμε τις αξίες μας. Ανησυχούμε για τις αυταρχικές τάσεις της Ρωσίας, ειδικότερα όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς αναφέρουμε αυτές τις ανησυχίες και σε διμερείς ε, και σε διεθνεί οργανισμού. Μίλησα με τον Μπόρι Τζόνσον την Παρασκευή, εξέφρασα την υποστήριξή μα και την αλληλεγγύη μα μετά από τι επιθέσει στο Σόλισμπορ. Ενθαρρύνουμε την Ρωσία να απαντήσει τι ερωτήσει που θέτει το Ηνωμένο Βασίλειο και ω απάντηση τη παραβίαση του διεθνού δικαίου από τη Ρωσία στην Ουκρανία, εμεί ε, μένουμε στο πλευρό των συμμάχων μα. Τα περιοριστικά μέτρα τη Νορβηγία ε, συνάδουν με αυτά ευθυγραμμίζονται με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πακέτο υποστήριξης ε, της Νορβηγίας ε, για την Ουκρανία ανέκτησε 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και για να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες παρέχουμε μεγάλη ανθρωπιστική υποστήριξη και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή την υποστήριξη και οικονομικά. Να πω και δύο λόγια για το Brexit, το οποίο δεν θα αλλάξει τη σχέση της Νορβηγίας με την Ένωση και αυτό το επαναλαμβάνω πολύ συχνά και στην Νορβηγία, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι θα συνειδητοποιήσουν ότι η σχέση μας παραμένει η ίδια. Εκτιμούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο υπογραμμίζει την ειδική, το ειδικό καθεστώς των συμφωνιών ε, ΕΖΕΣ και ΕΟΧ και βεβαίως ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός. Θέλουμε να διατηρήσουμε στενή σχέση και το κλειδί είναι η Συμφωνία ε, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που μας δίνει πρόσβαση στην ενιαία αγορά και εθώς και το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο όπως και για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Εξακολουθεί να παρέχει σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για τις οικονομικές σχέσεις της Νορβηγίας με τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Μέσω της, ε, του ΕΟΧ και των ε, νορβηγικών χορηγιών δίνουμε, προσφέρουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και, ε, μειώνονται έτσι οι κοινωνικές ανισότητες στα κρατη μέλη. Συμβάλλουμε και συνεργαζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ε, μαζί με τους, τα άλλα κράτη, ΕΟΧ και ΕΖΕΣ, δεν είμαστε απλές τρίτες χώρες σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που θα αλλάξει ωστόσο το Brexit θα είναι το νομικό πλαίσιο για την οικονομική μας συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία που επετεύθη ανάμεσα στους διαπραγματευτές Μπαρνιέ και Ντέιβις εχθές είναι μια θετική εξέλιξη, μια τακτική επόσυση και ένα νέο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις είναι σημαντικές για τις σχέσεις με την Ένωση βέβαια αλλά και με την Νορβηγία. Ε, και το τελευταίο μου παρατηρήση αφορά τις καθημερινές εργασίες της Επιτροπής κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιμετωπίζουν παρόμοιες ε, απειλέ ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο και σημαίνει αυτό αδιάκοπτη συνεργασία στην άμυνα και στι εξωτερικέ υποθέσεις, πράγμα που περιλαμβάνει και την Νορβηγία και τις χώρες του ΕΟΧ. Θέλουμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για στενές διαβουλεύσεις με χώρες που έχουν παρόμοιες απόψεις όπως εμείς. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η Ένωση θέλει να αυξήσει τις δυνατότητές της για να μπορεί να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις. Αυτό θα ενισχύσει ε, την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση και την αρβηγική ασφάλεια και είναι προς το συμφέρον της Νορβηγίας να συνεργαστεί στενά με την Ένωση και τα κράτη της Ένωσης στον τομέα αυτό. Είναι λοιπόν ουσιώδες να βρεθεί σωστός τρόπος ε, συνεργασίας στο ΝΑΤΟ και την Ένωση. Και επειδή ήμουν ε, υπουργό Άμυνα ε, με τον εδώ και τέσσερα χρόνια, να πω ότι η συνεργασία με την Νορβηγία είναι καλύτερη από ποτέ. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Θέλουμε λοιπόν βαθιά και ε, στενή σχέση με την Ένωση. Εμείς ε, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε ε, τις προκλήσεις στον κόσμο και στην άμεση μας γειτονία ως στενότεροι εταίροι και γείτονες. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ, για την παρουσίασή σας. Τώρα έχουμε χρόνια συζήτηση, πάνω από μισή ώρα, λίγο παραπάνω. Θα σας ενημερώσω αρχικά ότι σήμερα το πρωί το Διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε ότι θα μεταβούμε στην όμορφη σας χώρα τον Αύγουστο σε κοινή αποστολή των της Επιτροπής ΑΦΕΤ και της Υποεπιτροπής μας για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Θα πάμε στο Όσλο και μετά πολύ βόρεια. Βέβαια, βασικό στοιχείο είναι η ασφάλεια και η συνεργασία μας για την ασφάλεια. και όλοι οι συνάδελφοι περισσότερο ασχολούμαστε με το Brexit και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συχνά χρησιμοποιούμε την έκφραση το νορβηγικό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς οι Βρετανοί δεν θέλουν να ακολουθήσουν και είναι λάθο αυτή η απόφαση. Πολλά τα θέματα που θίξατε και πολλοί συνάδελφοι θέλουν να σας κάνουν ερωτήσεις. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πρώτος ο Μιχέλ Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω και εγώ θερμά στην Επιτροπή μας. Αν δεν ήξερα ότι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Νορβηγία, ακούγοντά σας μόνο, θα θεωρούσα ότι είστε καλό μέλος και πολύ καλύτερο από κάποια πλήρη μέλη. Εν πάση περιπτώσει, ε, αναφερθήκατε στα θέματα μέχρι στιγμής για το Brexit ε, φαίνεται να είστε ικανοποιημένοι από το τρόπο που βρισκόμαστε. Ξέρουμε ότι η Νορβηγία περιμένει εναγωνίως να δει τις εξελίξεις. Ε, γιατί είναι μέλος του ΕΟΧ, ε, ξέρω ότι δεν θα πει ποτέ ότι κοιτάξτε δεν είμαστε μέλος αλλά ε, και, και η Βρετανία τώρα που φεύγει έχει καλύτερη μεταχείριση από εμά. έχουμε υπόψη μας και ξέρω ότι τα έχετε κι εσείς. Μια ερώτηση, γιατί αναφερθήκατε στην Ακτική και τη συνεργασία με τη Ρωσία εκεί. Αν συγκρίνετε τη συνεργασία στο Συμβούλιο της Ακτικής φέτος ή πέρσι ή πρόπερσι, τι τύπος έχετε. Θεωρείτε ότι η Ρωσία θέλει να χρησιμοποιήσει το Συμβούλιο της ε, ε, Ακτικής για να ε, επιδείξει μια συμπεριφορά πάγια όπως είχε στο παρελθόν. Είναι πιο διστακτική, είναι πιο επιθετική, έχει αλλάξει η συμπεριφορά της. Και πέρα από το Ακτικό Συμβούλιο, στην ίδια την περιοχή υπάρχει στρατιωτική παρουσία, αυξάνεται. Πώς το εκτιμάτε εσείς. Φυσικά έχουν το δικαίωμα, όπως όλοι, να είναι παρόντες στο Σπίτσπερκ για λόγους ε, επιστημονικούς. Μόνο επιστημονική έρευνα κάνουν και κάνουν και τίποτα άλλο, κατασκοπία, ξέρω εγώ. Ε, φοβάστε. Ε, on, on, uh, Και σε σχέση με τις διμερείς σας σχέσεις, δεν απατώμε, έγινε ένα επεισόδιο όταν ήρθαν οι πρόσφυγες οργανωμένα ε, με ποδήλατα ε, από τους Ρώσους και φτάσανε στο Κίρκεμις. Έχετε συμφωνήσει με τους Ρώσους για να αποτρέπονται τέτοιου είδους ε, εχθρικά θέματα στο μέλλον ή πιστεύετε ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντάτε μία-μία τις ερωτήσεις. Όχι, να τις ομαδοποιήσουμε. Καλώς. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ο συνάδελφος κύριος Χάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ. Έχω ζήσει πολύ στην ωραία σας χώρα, όταν ήμουν νεότερος, ένα διάστημα. Θα ήθελα να σας ερωτήσω. Ε, έχετε συζητήσει με τον Υπουργό μας εξωτερικών ε, για το θέμα του Σάλτσμπερι. Εκφράσατε την αλληλεγγύη σας. Για το Brexit συζητήσατε με τον Υπουργό Εξωτερικών μας. Εγώ είμαι αναφανδόν υπέρ της παραμονής ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Θεωρώ τεράστια καταστροφή το Brexit, αλλά τι να κάνουμε εδώ. Πώς ε, βλέπετε το Ηνωμένο Βασίλειο να εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το έχετε συζητήσει με τον κύριο Τζόνσον. Και τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που παρετήθηκε. Τι λέτε για τα σχόλιά της και πώς εντάσσονται στην εξωτερική πολιτική. Μετά αυτή τη φοβερή επίθεση του, ε, του στη στην Νορβηγία, ε, τι γίνεται με την ε, συνοχή της νορβηγικής κοινωνίας. Και τέλος, Πολλοί Νορβηγοί έρχονται και μου μιλούν για κάποιους ε, ε, γάμους μεταξύ ε, ξαδέλφων που ακυρώνονται. Για ποιο νόμο μιλάτε? Ναι, είναι κάποιος νόμος για γάμους. Λίγο πιο αργά και λίγο πιο δυνατά μιλάτε. Παντρεύονται ξαδέλφια μεταξύ τους. Cousin marriages. Παντρεύονται ξαδέλφια. Ναι, και τώρα ακυρώνονται αυτοί οι γάμοι, από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλο θέμα και μου το έχουν θέσει πολύ υπόψη. Απέχει λίγο από το δικό σας χαρτοφυλάκι αυτό, αλλά θα πάρει καμία απόφαση η κυβέρνησή σας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Γιάννα Φωτίγκα. Madam, uh, welcome. Αγαπητή κυρία, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Σίγουρα είναι σημαντικό ο ρόλο τη Νορβηγία, το αναγνωρίζουμε τόσο σε θέματα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε θέματα συνεργασία στον τομέα τη ε, πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Συχνά φιλοξενούμε εκπροσώπου τη Νορβηγία και είμαστε σε διαρκή επαφή Θα ήθελα να συγχαρώ την Νορβηγία για τη συνεργασία της μαζί μας σε πολλούς τομείς. Στις σημερινές συζητήσεις ε, περί συνεργασίας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στον τομέα της άμυνας ε, και της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικές και οι δικές σας απόψεις. όλες οι παρατηρήσεις, ειδικότερα της Νορβηγίας και ειδικότερα μετά από τη Σύνοδο της Βαρσοβίας. Έχω κι εγώ μια ερώτηση για την Αρκτική. Όπως και ο συνάδελφος, αλλά θέλω να διευρύνω λίγο την ερώτηση. Θέλω να μου πείτε, από άψη στρατιωτικοποίησης της Αρκτικής, αλλά αν δούμε και λίγο πιο κάτω έχουμε το Καλίνιγκραντ που αμαυρώνει τις ελπίδες μας για μια ειρηνευτική διαδικασία στη Βαλτική. Και παρατηρούμε ότι και μετά από την προσάρτηση της Κρεμαίας ε, φοβόμαστε για την περιοχή του Καλίνιγκραντ ε, που στρατιωτικοποιείται και μετά ίσως και πιο νότια στη Μέση Ανατολή βλέπουμε άλλα προβλήματα. Τι πιθανότητες πιστεύετε υπάρχουν ε, να υλοποιηθεί το ψήφισμα 2401 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ώστε να υπάρξει γρήγορα και χειρία στη Συρία. Επίσης, ε, αναγνωρίζοντας ε, τον θετικό σημαντικό, σημαντικό ρόλο σας ε, στην ειρηνευτική διαδικασία της ε, Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας ε, για τα θέματα παιδείας στην Παλαιστίνη. Και τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών και πώς θα γίνει να αποφύγουμε τα ε, ακραίες περιπτώσεις στην Παλαιστίνη. Ευχαριστούμε κυρία και κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω στα σουηδικά στην ε, συνάδελφα από την Νορβηγία. Πρέπει να σας μιλήσω λοιπόν σουηδικά. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά την Αρκτική. Όπως είπατε κι εσείς, ε, έχουμε το θέμα της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής. Είναι καταστρεπτικές ε, οι συνέπειες ε, για μας που ζούμε στον Βορρά, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Ίσως ακόμη περισσότερο για άλλα μέρη του κόσμου. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου η Νορβηγία έχει πετρέλαια εκεί πάνω. Η εξόρυξη από βαθέα υδατά λοιπόν είναι κάτι αμφισβητήσιμο, είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, ακριβό και από όσο ξέρω έχει υπάρξει μια απόφαση του δικαστηρίου κατά ενός οργανισμού ε, ο οποίος ε, κατέφυγε στο δικαστήριο εναντίον της εξόρυξης ε, βαθαίων υδάτων. Οπότε, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την, ε, την Αρκτική, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πετρέλαιο θα παραμείνει εκεί που είναι. Έγινε και μια μελέτη στην Νορβηγία που έδειξε ότι πολλοί Νορβηγοί λένε ότι το πετρέλαιο δεν πρέπει να φύγει από εκεί που βρίσκεται, μέσα στο υπέδαφος. Πού βρισκόμαστε λοιπόν όσον αφορά την εξόρυξη πετρελαίου στην Αρκτική δεδομένων των σημαντικών συνεπειών που μπορεί να είχε κάτι τέτοιο. Έχουμε δει με αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο ότι είναι και στον κόλπο του Μεξικού είναι αδύνατο να περιορίσει κανείς ε, ένα ατύχημα εφόσον συμβεί. Επίσης αναφέρατε το Αφρίν. Χαίρομαι που το θέσατε. Είδαμε τι συνέβη πρόσφατα εκεί. αλλά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ε, μείνει εκοφαντικά σιωπηλές. Βλέπουμε να εμπλέκεται μια χώρα του ΝΑΤΟ, μια υποψήφια χώρα και υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά κανείς δεν λέει τίποτα, κανείς δεν καταδικάζει την κατάσταση, κανείς δεν καταδικάζει τα όσα κάνει η Τουρκία. Η Νορβηγία έχει μια πιο ευέλικτη θέση, μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά από τους υπόλοιπους εμάς. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι λέει η Νορβηγία για την κατάσταση αυτή και τι σχεδιάζει να κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ms. We have two more speakers. Ευχαριστώ κυρία Βαλέρο. Έχουμε δύο ακόμα ομιλητέ. Επόμενο είναι πρώην Πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών, ο κύριο Έλμαρ Μπρόκ από τη Γερμανία. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Θυμάμαι τις συζητήσεις που είχαμε στο Όσλο πριν από μερικά χρόνια. Uh, και θέλω να ρωτήσω κάτι ε, για την πολιτική ασφαλεία σε συνδυασμό με το Brexit. Θα πρέπει να βρούμε μια ειδική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και για τα θέματα ασφαλείας, ιδιαίτερα μετά την ΠΕΣΚΟ, την μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και πώς μπορούμε να προσκαλέσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να παίρνει μέρος σε ε, αποστολές, δημόσιες προμήθειες, συμβάσεις ε, μυντικές κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε. Γιατί αντίστοιχες καταστάσεις γνωρίζετε. Πώς μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια δραστηριότητα μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που είναι η Νορβηγία, που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά δεν μπορείτε να συμμετέχετε στη διακυβέρνηση, αλλά με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η σύνθεση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, και ο Πρωθυπουργός είπε πριν από λίγο καιρό ότι στη διαπραγμάτευση του Brexit, αν δεν θέλει το Ενωμένο Βασίλειο να ε, έχει τη συμμετοχή της Νορβηγίας στην εσωτερική αγορά που δεν είναι μέλος, δεν μπορεί να είναι σε καλύτερη μοίρα το Ηνωμένο Βασίλειο από την Νορβηγία και να έχει καλύτερη μεταχείριση. Θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά πράγματα σχετικά. Ευχαριστώ, Έλμα. Και τέλος, ο κύριος Πέτερλε από τη Σλοβενία. Γεια σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ για τα σαφή και φιλικά σας λόγια. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, το εξής. Πρόσφατα ρώτησα ένα πολιτικό φίλο μου από μια χώρα που είναι πιο κοντά στη Βρυξέλλες από την Ορβηγία. Τι θεωρούν για την Ουκρανία στη χώρα μου σου. Και μου λέει, μα η Ουκρανία είναι τόσο μακριά άλλο από εμά. Και χαίρομαι που για την Νορβηγία Τίποτα δεν θεωρείται μακριά, ούτε τα Δυτικά Βαλκάνια. Ακόμα και σε αυτά εστιάζετε την προσοχή σας και χαίρομαι ε, γι' αυτό. Είπατε ότι μοιραζόμαστε αξίες και γεωγραφία. Μακάρι να τα έλεγε και κάποιος άλλος όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Είστε έτοιμοι να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. Και ένα σχόλιο ε, από πλευρά μου. Εγώ πήγα ε, στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και τις επισκέφθηκα στη Λιθουανία πριν από λίγες εβδομάδες ε, το γερμανικό τάγμα στην Ούκλα και είναι και Νορβηγία εκεί ανεπτυγμένη. Εξαιρετική και πάλι συνεργασία. Είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Νορβηγία στο ΝΑΤΟ. Όπως είπε και κάποιος συνάδελφος μόλις. Ακούγοντάς σας, φαίνεται ότι η Νορβηγία είναι καλύτερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κάποια νυν μέλη, περιπτώσει. Ε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις. Ε, καταρχάς, ε, με χαρά θα σας καλωσορίσουμε στην Ολυμπιακή τον Αύγουστο. Είναι πολύ καλό ε, χρόνο. Πολύ χρονικό, καλό χρονικό διάστημα. Έχουμε λοιπόν πολύ καλή συνεργασία με χώρες όπως η Λιθουανία αυτή τη στιγμή όπου είμαστε πλάι-πλάι όπως έχουμε κάνει στη Διεθνή Φόρα εδώ και δεκαετίες και αυτό είναι κάτι που καθιστά τη συνεργασία μας ακόμα βαθύτερη και ε, Πιστεύουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή επιτείνει τις προσπάθειες με την ε, την ΠΕΣΚΟ για παράδειγμα, ε, με τη μόνιμη διαστομένη συνεργασία, είναι θέμα ασφάλειας ολονών και αυτό ακριβώς κάνουμε. Υποστηρίζουμε με τους ΔΕ, αυτό είναι το ΝΑΤΟ και η ΟΗΕ, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, ε, για να μπορούμε να σταθούμε ε, και αν δεν το κάναμε δεν θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και στις διεθνείς, στους διεθνείς οργανισμούς και να αλληλοπροστατευόμαστε. Νομίζω λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό το θέμα των αξιών. Πρώτη ερώτηση από Μίχαλ Γκάλερ για το Brexit και επίσης ε, το Συμβούλιο της Αρκτικής. Η εντύπωσή μου είναι πως η συνεργασία στο Συμβούλιο της Αρκτικής λειτουργεί καλά με όλες τις χώρες και όλους τους παρατηρητές που συμμετέχουν και έχει γίνει έτσι, έχει παραμείνει έτσι από το 2014 και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία. Ίσως ε, θα πρέπει, λέει, να ε, γίνουν δε συζητήσει για την ασφάλεια στο Συμβούλιο της Αρκτικής. Εγώ θα έλεγα πως όχι γιατί το Συμβούλιο της Αρτικής είναι ένας χώρος συνεργασίας για την περιφέρεια αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλές χώρες στις περιφέρειες να μείνουν στην ησυχία τους γιατί λειτουργεί έτσι πως είναι αυτός ο κύκλος, ε, αυτό το Συμβούλιο για την ώρα. Υπάρχουν άλλα φόρα που ασχολούνται με την ασφάλεια περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά την αυξημένη στατιωτική δραστηριότητα από τη Ρωσία στο βορρά, εμείς βλέπουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το άνοιγμα εκ νέου πολλών βάσεων που είχαν κλείσει για δεκαετίες ορισμένες. Ορισμένες εξ αυτών είναι για πολιτικούς σκοπούς, γιατί δεν υπάρχουν πολλές υποδομές στην περιφέρεια και αν θέλει κανείς απλά και μόνο να κάνει μια εξερεύνηση, θα πρέπει να έχει κάποιες ε, σταθερές υποδομές. Υπάρχουν όμω και άλλε που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικού καθαρά σκοπού. Κάτι ακόμα που βλέπουμε είναι αυξημένη δραστηριότητα και ένα συγκεκριμένο σχήμα δραστηριότητα. Βλέπουμε δηλαδή σε πολλούς τομείς, σε πολλές περιοχές, όχι απαραίτητο στο βορρά, αλλά α πούμε και στη Βαλτική θάλασσα, πιο επιθετική συμπεριφορά. Βλέπουμε περισσότερο, πιο περίπλοκα σχήματα πτήσεων, αυξημένη παρουσία, θαλάσσια παρουσία, αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι μόνο στρατιωτικά τα μέσα. Βλέπουμε και αυξημένη δραστηριότητα όσον αφορά την προπαγάνδα και τα μηνύματα. Υπάρχει δηλαδή κατασκοπία, μεγάλη δραστηριότητα κατασκοπική η κοινότητα κατασκοπική ε, τελευταία φορά μας έδωσε ενημέρωση στις 6 Μαρτίου όπου μας έδωσαν μια πολύ ειλικρινή ακτίμηση του γεγονότος ότι η Ρωσία και η Κίνα μας δημιουργούν προβλήματα και προκλήσεις όσον αφορά την κατασκοπία. Εμάς και σε άλλες χώρες όμως. Τώρα, Ηνωμένο Βασίλειο να μπει στον ΕΟΧ, ρωτήσατε. Μέχρι στιγμής δεν είναι στην ατζέντα αυτό το θέμα. Λόγω των αποφάσεων που λήφθησαν στην ίδια την Βρετανία. Και όταν ακούει κανεί την Τερέζα Μέη και ακούει την ομιλία τη στις 2 Μαρτίου, ήταν σαφές ότι η εσωτερική αγορά και η τελωνιακή αγορά θα η τελωνιακή ένωση θα μείνουν. Άρα είναι απαραίτητε προποθέσει αυτά. Κατά τη γνώμη μας η ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντική, γιατί έτσι έχουμε πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά μισούδης ανθρώπων για όλες τις επιχειρήσεις και για όσον αφορά την προβλεψιμότητα της οικονομικής μας ισχύω. Είναι εσωτική σημασία. 80% των εξαγωγών μας ε, πηγαίνουν στην Ένωση. Και βεβαίως ε, πολύ θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς μας σημαίνει πολλά για μας και πολλά και για τις χώρες τις υπόλοιπες του ΕΟΧ. Είναι ένα θέμα λοιπόν που δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις. Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και καιρό όσον αφορά τους γάμους μεταξύ εξαδέρφων. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ όχι μόνο την Νορβηγία αλλά και τις άλλες χώρες όπου συζητείται το θέμα, αλλά ακόμα αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Τώρα, για το θέμα της συνεργασίας με την ΚΕΠΑ και την... το ΝΑΤΟ. Κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και ΝΑΤΟ και τις ρωσικές δραστηριότητες, στρατιωτικές δραστηριότητες όσον αφορά την ε, εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν με εντυπωσιάζει και πολύ πως είναι πολύ δύσκολο να επιβληθούν αυτά τα ψηφίσματα διότι ε, πρέπει να υπάρξει πάυση του πυρός από όλες τις πλευρές. Ε, ε, Για την ώρα οι ανακοχές έχουν διαρκέσει μόνο κάποιες ώρες και μόνο πολύ λίγοι διάδρομοι έχουν ε, ε, ε, λειτουργήσει όπου έχει κενωθεί η χώρα. Μου είπαν ότι έχουν γίνει 50 μεταγωγές ιατρικού τύπου ενώ χρειάζονται πολύ περισσότερες, κυρίως γυναίκες και παιδιά είναι μπλοκαρισμένα στους διαδρόμους από την Κούτα. Είναι πήγουσα κατάσταση. Πρέπει λοιπόν με ισχυρή φωνή να ζητήσουμε από τα μέρη να σεβαστούν αυτό το ψήφισμα. Να γίνει ανακοχή ώστε να ανακουφιστούν οι άνθρωποι επιτόπου. Η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ε, το θέμα της παιδείας. Σε αυτό το θέμα συνεργαζόμαστε πολύ με την ΟΝΡΑ. Ε, έχουμε την αξιολόγηση των, της ύλη για την πρώτη τάξη μέχρι την τελευταία του Δημοτικού και τώρα κοιτάμε τις υπόλοιπε γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε για τα μικρότερα παιδιά αυτά που πάνε σχολείο δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο μεθαρρύνουμε. Ε, ξαφνικά έχασα τη λέξη που έπρεπε να πω. Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς να ενθαρρύνουμε οποιοδήποτε είδος ε, μηνυμάτων μίσους ε, μεταξύ τους. Γιατί αν τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν μέσα στο μίσος, ε, τότε η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να βρεθεί μια διαρκής ειρήνη στην περιοχή και να διατηρηθεί. Αρκτικός κύκλος. Ε, αυτό που μπορούμε να πούμε για τις κλιματικές αλλαγές στην Αρκτική θα πρέπει να πούμε ότι επηρεάζει την Αρκτική, αλλά δεν προκύπτει από την Αρκτική. Απλά φαίνονται πολύ γρήγορα οι επιπτώσεις στην Αρκτική. Γι' αυτό και είναι ένα τεράστιο εργαστήριο για να δούμε, να ερευνήσουμε και να βρούμε τρόπους πρόβλεψης για το τι θα γίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Όπως γνωρίζετε από το 1979 κάνουμε μια κάνουμε εκμετάλλευση φυσικού αερίου και πετρελαίου φιλικού προς το περιβάλλον. Ε, υπάρχουν περιοχές που δεν είναι ανοιχτές στην εξόριξη, ακριβώς επειδή είναι πολύ ευάλωτες, αλλά το, το κάνουμε αυτό και όταν όντω κάνουμε εξόριξη πετρελαίου ή φυσικαριού, το κάνουμε με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και θέλουμε να συνεχίσουμε. Είναι σημαντικό οτιδήποτε κάνουμε όσον αφορά την εξόριξη φυσικών πόρων, ιδιαίτερα των μη ανανεώσιμων, Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι, ότι δεν θα συμβούν ατυχήματα και ότι το περιβάλλον και ε, γύρω περιοχές δεν θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι αυτό που είναι ανεκτό για το περιβάλλον. Um... τώρα. Μίλησα για την εξωτερική πολιτική στο Κοινοβούλιο. Κάθε χρόνο το κάνω αυτό. Και ήταν σαφές το μήνυμα ότι εγώ και η νορβηγική κυβέρνηση ανησυχούμε πάρα πολύ για το επίπεδο δραστηριότητας της Τουρκίας. Επίσης ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσουμε σε όλα τα μέρη ότι υπάρχουν κανόνες μεταξύ άλλων για την αναλογικότητα που πρέπει να τηρηθούν για να είμαστε και σύμφωνοι με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Αυτό που κάνουν κάποιες χώρες ε, για παροτρύνουν στην προσοχή και στην αυτοσυγκράτηση είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις στην περιοχή για πάρα πολύ καιρό και υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Όλα πρέπει να γίνουν με αναλογικό τρόπο. Η κλιμάκωση που είδαμε τις τελευταίες μέρες μας κάνει να ανησυχούμε περισσότερο και μόνο το τελευταίες τρεις-τέσσερις μέρες η κλιμάκωση ήταν ε, ε, πολύ μεγάλη. μάρα. Νομίζω πως η συνεργασία με την ε, συνεργασία ε, την ΠΕΣΚΟ και ε, είμαστε συνδεδεμένοι με την Οργανισμό Άμυνας εδώ και πολλά χρόνια και είμαστε ο 7 μεγαλύτερο μεγαλύτερος ε, συνεισφέρον. Όμως θα θέλαμε να βρούμε τρόπους για project μονομένα project στο ΠΕΣΚΟ Είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς τι είδους συνεργασία έχουμε. Αλλά ούτως ή άλλως και πριν την ΠΕΣΚΟ, εμεί αναζητούσαμε τρόπους για στενότερη συνεργασία. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι θα πρέπει να βρούμε επιπλέον ε, τρόπους συνεργασίας χωρίς να επικαλύπτονται όμως οι δομές και οι δραστηριότητες. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δούμε ποια πράγματα θα κάνει καλύτερα το ΝΑΤΟ, ποια πράγματα θα κάνει καλύτερα η Ένωση, ώστε να φροντίσουμε καλύτερα γενικά την ασφάλειά μας. Έχω μιλήσει και με την Κομισιόν ε, ΔΕ για τη συμμετοχή μας στην προπαρασκευαστική δράση για την αμυντική έρευνα. Συμμετέχουμε, νομίζω πως είμαστε η μόνη τρίτη χώρα που συμμετέχει μέσω του ΕΟΧ. Αλλά για την αμυντική μας βιομηχανία είναι σημαντικό να συμμετέχουμε και στο βιομηχανικό πρόγραμμα, γιατί θα έχουμε πολλούς πόρους που θα πάνε στην έρευνα. Και βεβαίως για να ωφεληθούμε από αυτό θα πρέπει θα πρέπει να είμαστε μέρο του προγράμματο του βιομηχανικού. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα. Μιλάμε με μονομένα με χώρε, μιλάμε με την Κομισιόν για να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, και αξιόλογο και για την Ένωση να μας έχει τέρους αφού είμαστε μέρη στον ΕΟΧ και στην προπαρασκευαστική δράση. Τέλος. Τώρα, περισσότερο σχόλιο παρά ερώτηση όσον αφορά την Ουκρανία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που κάνουμε σε συνεργασία με την Ένωση, στο ΝΑΤΟ και διμερώς με την Ουκρανία, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε την διαδικασία μεταρρύθμισης ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Ουκρανία είναι πράγματα που προσπαθούμε να διορθώσουμε με την, την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να σταθούμε και να επιμείνουμε στις αξίες μας. Αν και έχω καταγράψει πολλές φορές ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κόπωση από πλευρά της Ουκρανίας, ότι δηλαδή ε, θα, ε, εμείς θα πρέπει να μείνουμε σταθεροί και να δίνουμε πάντα το ίδιο ξεκάθαρο μήνυμα. Πρόκειται για ρήξη του διεθνούς δικαίου και γι' αυτό και έχουμε να πάρει μέτρα και γι' αυτό και στηρίζουμε την Ουκρανία σε αυτή την τόσο δύσκολη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ε, άλλες ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις έχετε. Όχι. Άρα, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά που ήρθατε. Καλή συνέχεια. Ε, έχετε μια επιτυχή μέρα στη Βρυξέλλες. Ακούσαμε σήμερα το πρωί ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και συναρπαστική η πολιτική κατάσταση Ε, στη Νορβηγία. Φτάνοντα στι Βρυξέλλε, δεν ξέρατε αν έχει πέσει η κυβέρνησή σα ή αν έχει αντέξει την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Ήταν εξαιρετική πάντω η ανταλλαγή απόψεων με όλη την Επιτροπή και σα ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Εγώ σα ευχαριστώ που με καλέσατε. So, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζεται τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρώτο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας του Κωσυφοπεδίου, τον κύριο Μπέτζετ Πατσόλη. Ελπίζω σωστά να το... ή Πατσόλη. Πατσόλη μάλλον. Ο κύριος Μπέτζετ Πατσόλη λοιπόν Καλωσορίσατε, Υπουργέ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι χαρά και τιμή μας να σας υποδεχόμαστε. Βεβαίω θέλω να καλωσορίσω και τον πρέσβη του Γοσφοπεδίου ε, στις Βρυξέλλε, τον Μπέρνατ Νίκαη, ο οποίος είναι τακτικός επισκέπτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπουργέ, εισαγωγικά, τα Δυτικά Βαλκάνια καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα της καθημερινής μας δουλειάς εδώ. Μερικοί συνάδελφοι και ο εισηγητής ο Ίγκο Σόλτες, αλλά όχι μόνο, ασχολούμαστε περισσότερο ε, με τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τι δείχνει αυτό, όχι απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αποδίνουν πολύ μεγάλη σημασία στη διαδικασία μετάβασης και μετασχηματισμό της περιοχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ε, στη διαδικασία ένταξης και των έξι κρατών. Βέβαια, ο καθένα θα κρίνεται με βάση τις επιδόσεις του. Το κοσφοπέδιο είναι τμήμα της διαδικασίας διεύρυνσης και το υποστηρίζουμε στο δρόμο και στην πορεία του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργέ. Η στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες εβδομάδες, κατά την άποψή μου στέλνει ένα νυφάλιο μήνυμα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για να επέλθουν γενικά στην περιοχή και ειδικά στο Κωσυβοπαίδιο θετικές αλλαγές. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Και μάθαμε ότι προέρχηση από τον ιδιωτικό τομέα ξέρετε τα πράγματα και μας τα λένε και κοσοβάροι ε, γνωστοί αυτά και ξέρετε από τον ιδιωτικό τομέα ότι χρειάζεται καμιά φορά και στην πολιτική ε, να γίνονται συμβιβασμοί και, και, στην πολιτική θέλουμε εταίρους ε, αυθεντικούς, γνήσιους, ειλικρινείς και αξιόπιστους θα σας δώσω το λόγο για να μας μιλήσετε για τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σας και τι βοήθεια χρειάζεται και υποστήριξη για να γίνουν τα απαραίτητα. Φαντάζομαι οι συνάδελφοί θα ενδιαφερθούν να ακούσουν ιδιαίτερα τις απόψεις σας για το μη κλειδιά όπως είναι. Ε, τα τελικά βήματα για την απελευθέρωση θεώρησης ε, διαβατηρίων το είδαμε το αντίστοιχο με το Μαυροβούνιο. Το δεύτερο μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της ζωσπαστικοποίησης και του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα σας. Και τέλος, χωρίς αυτό να είναι το λιγότερο σημαντικό, δικαιοσύνη και συμφιλίωση. Με πλήρη συνεργασία και φυσικά με τα, τους αρμόδιους φορείς και αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι και ο διάλογος Πρίστινας Βελιγραδίου. Πολύ σημαντικά τα θέματα και πάλι με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε. Έχετε το λόγο, Υπουργέ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Αποτελεί τιμή για μένα να απευθύνω το λόγο σε αυτό το τόσο σημαντικό ακροατήριο. Την ομιλία μου την έχω γραπτός και θα τη διαβάσω Έχω και μερικέ λέξει στα ισπανικά και μερικέ στα γερμανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι τη Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη μου τιμή που έχω την ευκαιρία να σα απευθύνω το λόγο σήμερα. Θα ήθελα να εκφράσω πρώτα απ' όλα την εκτίμησή μου και το βαθύ σεβασμό και τις ευχαριστίες ε, της χώρας μου για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να υπογραμμιστεί ρητά ότι το μέλλον της δημοκρατίας του Κωσυφοπεδίου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από την ε, διακήρυξη της ανεξαρτησίας, η ολοκλήρωση, στην Ευρωπαϊ... η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ είναι η βασικότερη στόχοι της κοινωνίας μας. Είμαστε περήφανοι που έχουμε παγιώσει αυτές τις αρχές ε, που διέπονται από το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Η νόμη μας, ε, ε, το σύνταγμά μας, η διακυβέρνησή μας είναι κατ' ουσίαν ευρωπαϊκέ. Ευρωπαϊκές είναι οι αξίες που διέπουν την κοινωνία μας και τη χώρα την οποία οικοδομήσαμε μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Ε, σύμφωνο απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεσμευόμαστε με τις ίδιες δεσμεύσεις ε, της εργασίας σας στο Στρασβούργο, τα σημαντικά ψηφίσματα, τις ανταλλαγές ε, και τη βοήθεια που μας παρέχετε πρακτικά από τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το, η υπηρεσία, το ULEX, της ε, αντιπροσωπής των κρατών μελών. Είναι σημαντική η συμβολή τους, γι' αυτό θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του Κωσυφοπηδίου. Σας κάνω έκκληση να συνεχίσετε τη δέσμευσή σας, ε, να μας βοηθάτε, όπως και την υπόλοιπη περιοχή ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα, ειρηνική ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια. Κάτι που θα έχει θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή εμείς στα Δυτικά Βαλκάνια βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη εποχή ε, της ευρωπαϊκής μας διαδρομής. Έχει δημοσιευτεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και στη συνέχεια είχαμε την ομιλία του δήλωση του κυρίου Γιούνκερ και τη κυρία Μογκερίνη και του κυρίου Χάν, οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή, αυτό έδειξε τη σαφή δέσμευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά και τα κράτη-μέλη εντείνουν την δέσμευσή του στην περιοχή. Η Βουλγαρική Προεδρία κατέστησε τα Δυτικά Βαλκάνια μια βασική προτεραιότητα στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφή στη Σόφια για τα Δυτικά Βαλκάνια και η διαδικασία του Βερολίνου και η διασκέψη του Λονδίνου. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι Υπάρχει ένα σημαντικό μήνυμα ότι οι κάτοικοι των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να αντιληφθούν ότι η χώρα έχει μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή προοπτική. Πρέπει να υποθεί ότι στο κοσυφοπαίδιο η αξιοπιστή αυτή της προοπτικής συνδέεται άρρηκτα με την απελευθέρωση. Πριν προχωρήσω, ήθελα να μιλήσω για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήματα ε, στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Οι πολίτες μας είναι η μόνη της περιοχής που ακόμα δεν ε, εντάσσονται σε κάποιο καθεστώς ε, απαλλαγής θεωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε νεαρό πληθυσμό, εκπαιδευμένο, γεμάτο ενθουσιασμό για κάθε τομέα, αλλά σήμερα αισθάνονται απομονωμένοι. Για αυτούς είναι δύσκολο να αντιληφθούν, να καταλάβουν πώς θα προχωρήσουν προς τα μπρος τους λείπει το βασικό δικαίωμα ε, επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επιλύσουμε το παρόν πρόβλημα επιγόντως. Ας δούμε δύο προϋποθέσεις, ε, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτον την κύρωση των συνόρων με το Μαυροβούνιο. Το Κωσυφοπέδιο έχει κάνει ό,τι μπορεί για να καταλήξουμε σε κάποιο σε κάποια κατάληξη. Ε, είχαμε δυστυχείς εσωτερικές πολιτικές επιπλοκές, αλλά βρισκόμαστε στο τέλος ε, της διαδρομής και σήμερα η συνέλευση του Κωσφοπεδίου θα συναντηθεί και ελπίζουμε ότι θα κυρώσει το σύνορα με το Μαυροβούνιο. Με το Μαυροβούνιο μάλιστα ξέρετε έχουμε άριστες ε, σχέσεις, σας το λέω ενημερωτικά. Πρέπει να ενισχύσουμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της ε, διαφθοράς. Εκεί έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Οι εργασίε αυτές γίνονται από το ανεξάρτητο δικαστικό σώμα και εμεί ω κυβέρνηση έχουμε διασφαλίσει να υπάρχουν απαραίτητες ικανότητες που θα δώσουν τη δυνατότητα να επιτύχουν αυτοί οι θεσμοί αποτελέσματα. Ταυτόχρονα έχουμε ενημερώσει ε, τις αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται επί τόπου και τη Βρυξέλλες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Αφού κυρωθεί ε, το όριο, το σύνορο, θα έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η δουλειά σε αυτό το τομέα δεν θα ολοκληρωθεί έτσι, αλλά είναι ένα σημαντικό στοιχείο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι την προσχώρηση και μετά από αυτήν. Ωστόσο, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, έχουμε επαρκείς προϋποθέσεις που πληρούνται για τους σκοπούς της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Έχουμε ένα μικρό αριθμό ετούντων άσυλο, ε, περίπου 7.000. Ε, αυτός ο μικρός αριθμός φέρνει το κοσυφοπέδιο πίσω από τις χώρες ε, της περιοχής που έχουν ε, θεωρήσει σήμερα η Αλβανία και η Σερβία σήμερα. Ε, έχουν ε, δημιουργηθεί η νομοθεσία και το πλαίσιο που απαιτούνται και τώρα υπάρχει ένα υφόρο σύστημα που δεν θα επιτρέψει περαιτέρω αύξηση στον αριθμό των παράτυπων μεταναστών ελπίζουμε ειλικρινά ότι μέσω της στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορέσουμε να παρέχουμε στους πολίτες μας ε, την ελευθερία κυκλοφορίας. Αν μπορείτε να κάνετε κάτι και εσείς φέτος για να μας βοηθήσετε, δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε το όνειρο αυτό του κοσυφοπηδίου πραγματικότητα, να νιώσουμε ίσοι με τους γείτονές μας, ε, να απολαμβάνουμε και εμείς ε, το ίδιο δικαίωμα με αυτούς. Θα, επιτρέψω, θα επιστρέψω τώρα στην ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο Κωσυφοπαίδιο μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης φέτος. Η θέση μας θα ενισχυθεί με τη νέα συμφωνία που θα επιτρέπει στο Κωσυφοπαίδιο να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα η στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια της Νέα Επιτροπής ε, δημιούργησε μια νέα δέσμευση όχι μόνο για την ευρωπαϊκή προοπτική ολόκληρης περιοχή, αλλά ενίσχυσε και την υποστήριξη που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη στρατηγική, ειδικότερα δεδομένη τη πολιτική πίεση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Να μην υποσχόμαστε υπερβολικά πολλά. και ώστε να επιτύχουμε το, να φέρουμε σε ζωή το όραμα της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ταυτόχρονα θα ήταν παράληψη να μην πω ότι αναμένουμε στο μέλλον να γίνει ακόμη πιο συγκεκριμένη η ευρωπαϊκή μας προοπτική. Το Κωσυφοπέδιο έχει μια σαφή φιλοδεξία να γίνει χώρα ε, υποψήφια ε, για μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης το συντομότερο δυνατόν. Αυτό αναμένει και ο λαός του Κωσυφοπεδίου. Αναμένει μια συγκεκριμένη προοπτική ευρωπαϊκής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίση μεταχείριση όλων των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό σημαίνει άρση των εμποδίων ε, στη συνδεσιμότητα στις οικονομικές ανταλλαγές ε, και, στην επίλυση, και επίλυση των διμερών πολιτικών ζητημάτων. Δυστυχώς μερικές φορές ε, ύπαρξη κάποιων ζητημάτων όχι απλά μας εμποδίζει να προχωρήσουμε αλλά δυστυχώς ε, μερικές φορές μας οδηγεί και σε ε, ε, υποχώρηση στις σκοτεινές πρακτικές του παρελθόντος. Είχαμε τις παρεμβάσεις της Σερβίας στις εσωτερικές μας υποθέσεις αλλά και, στις προσπάθειε και τις προσπάθειες υπονόμευσης της διεθνούς μας Μας εντείνουμε, βλέπουμε μια ε, όλο και πιο έντονη ε, εκστρατεία της ε, Σερβίας να πείσει χώρες που μας έχουν αναγνωρίσει να άρουν αυτή την αναγνώριση ή να αμφισβητήσει την ιδιότητα μέλους του κοσμοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς. Εδώ θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον διάλογο διευκόλυνση ε, τη ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Σερβία. Ο διάλογο έχει μπει στην τελευταία φάση στο Κωσυφοπαίδιο, έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση, καλόπιστη υλοποίηση όλων των συμφωνιών στην περιοχή και τη Συμφωνία σύνδεση των Δήμων ε, Σερβικής ε, πλειοψηφία ε, σύμφωνα με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κωσυφοπαιδίου και ελπίζουμε οι Σέρβοι ομολογοί μα να δείξουν επίσης τη θέληση να υλοποιήσουν τη συμφωνία για την ενέργεια και να αναγνωρίσουν τα διπλώματα και να σταματήσουν τις προσπάθειές τους να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του κοσφοπεδίου στην UNESCO, στην Interpol και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτή τη φάση του διαλόγου θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ώστε να μπορέσουμε και οι δύο χώρες να προχωρήσουν προς την Ευρώπη ε, και στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου ε, και προς το σύμφωνο, στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα για την οικονομία. Η οικονομία αναπτύσσεται στο Κωσυφοπεδίο κατά 4% τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας ε, και να χρησιμοποιήσουμε πιο βιώσιμους πόρους για την ανάπτυξη. Έχουμε σαφή βελτίωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο κοσφοπέδιο. Έχουμε ανέβει 20 θέσεις σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας μέσα σε ένα χρόνο. Πέρυσι μπορέσαμε να ανακοινώσουμε την υπογραφή μιας συμφωνίας ε, για μια από τις μεγαλύτερες άμεσες επενδύσεις ε, που έχουν γίνει σε ένα ε, εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής επενδύσαμε Είχαμε μια επένδυση στο κοσφοπέδιο δηλαδή ε, για την οικοδόμηση ενός ε, εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής ε, τέ, τέτοιας δυναμικότητας που ήταν μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο κοσφοπέδιο. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, πολλές δυνατότητες και αναμφίβολα το κοσυφοπέδιο έχει πολλές τέτοιες δυνατότητες, αλλά οι ευκαιρίες αυτές ε, δεν ε, αξιοποιούνται επαρκώς. Κάτι άλλο που θα μας βοηθήσει στην περιοχή θα είναι η μελλοντική οικονομική ολοκλήρωση. Είμαστε έξι αυτόνομες χώρες στην περιοχή, ανεξάρτητες χώρες ε, και είμαστε όλες ελεύθερες δημοκρατίες με οικονομίες αγοράς. Έχουμε όλες δυνατότητες ανάπτυξης αλλά τα διαρθρωτικά και πολιτικά εμπόδια που υπάρχουν ακόμα εμποδίζουν την οικονομική ολοκλήρωση. Θα πρέπει αυτά να επιληθούν ή να έρθουν για να μπορέσουμε τελικά να μιλήσουμε για μια πραγματική περιφερειακή, για ένα πραγματικό περιφερειακό οικονομικό χώρο. Εμείς είμαστε υπέρ της άρσης αυτών των εμποδίων για το εμπόριο. Είμαστε υπέρ μιας περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης γιατί πιστεύουμε ότι ε, οι στενότεροι περιφερειακοί οικονομικοί δεσμοί θα μας βοηθήσουν στο διαδρομή προς την ε, ε, Ευρώπη. Η οικονομική αλληλεξάρτηση επίσης θα συμβάλλει σε μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια συνεπώς για τους πολίτες μας. Θα διασφαλίσει συνδεσιμότητα σε όλη την περιοχή σταθερότητα και άριστες σχέσεις. Πιο ευρέως ε, έχουμε εστιαστεί στο να διασφαλίσουμε την ένταξη της χώρας μας ε, στη διεθνή κοινότητα. τόσο μέσω της συμμετοχής σε διεθνούς οργανισμούς όσο και μέσω της αναγνώρισης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 117 αναγνωρίσεις και συνεχίζουμε τις προσπαθίες μας. Φυσικά η αναγνώριση από τα πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μας έχουν αναγνωρίσει ακόμα είναι προτεραιότητά μας και λυπούμαστε που αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής ε, η στάση τους έχει επηρεαστεί από εγχώρια προβλήματα όσον αφορά την ανεξαρτησία μας. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν κατά επανάληψη και το επαναλαμβάνω το Κωσυφοπαίδιο είναι μια μοναδική χώρα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα ιστορικά Τέλος, θα πρέπει να πω ότι ε, κηρύξαμε την ανεξαρτησία μας γιατί ήταν η μόνη λύση για να επιβιώσουμε φυσικά στη γενοκτονία ε, που ε, υπέστη η ε, εθνότητά μας. Η ανεξαρτησία μας οφείλεται σε μοναδικές συγκυρίες ε, που μας οδήγησαν σε αυτό και είναι μη αναστρέψιμη. Χαιρόμαστε και είμαστε περήφανοι που μας έχουν αναγνωρίσει 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και οι πέντε εναπομείνασες χώρες, εάν μας ε, αναγνωρίσουν, ε, θα είναι πολύ ενισχυτικό για μας. Ε, δεν είναι μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας μας. Αγωνιστήκαμε μαζί με τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ, για να επιβληθεί ένας ε, νόμος διεθνής, μια απόφαση για την ανεξαρτησία. Άρα η ανεξαρτησία μας δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δικαστήριο Απεφάνθη άλλωστε επίσης ότι η ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου είναι sui generis. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προηγούμενο. Ο τροχός της ιστορίας δεν γυρίζει πίσω. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και μπρο για στο το κουσιφοπέδιο. Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε ε, στη δική μας διεθνή παρουσία και εδραίωση και βελτίωση της θέσης να έχουμε περισσότερες υπηρεσίες, περισσότερη απασχόληση, περισσότερες ευκαιρίες για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Άλλωστε αυτό περιμένουν και οι πολίτες. Βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, αναθεώρηση οικονομικής διακυβέρνησης ε, και πιο αποτελεσματικό κράτος δικαίου είναι οι προτεραιότητές μας. Σε αυτό το δρόμο επίσης θέλουμε να κλείσουμε και οποιαδήποτε διμερεί θέματα που εκκρεμούν και να ολοκληρώσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις για να βεβαιωθούμε ότι θα περάσουμε στο επόμενο βήμα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής μας ένταξης, λαμβάνοντας ε, το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή στο προσεχές μέλλον. Στο δρόμο μας λοιπόν για τις βασικές μεταρρυθμίσεις και για τη βελτίωση ε, των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών μας, μας ε, συνοδεύσατε σε κάθε βήμα μας, όπως και στην εκπλήρωση της βαθιάς μας επιθυμίας να γίνουμε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κόσοβο σας ευχαριστεί πολύ και στα Ιταλικά επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, συμπαράστασή σας και η πρόκληση συνεχίζεται. Για μας θα ήταν ένα βραβείο που πραγματικά αξίζει μια επιβράβευση του Κωσοφοπέδιου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια των Εθνών. Σας ευχαριστώ σε διάφορες γλώσσες. Ευχαριστούμε, Υπουργέ Πατσόλη. Και επίσης που απευθυνθείτε σε εμά σε διάφορες γλώσσες των κρατών μελών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και μας αρέσει αυτό. Και τώρα, έχουμε περίπου μισή ώρα για ανταλλαγή απόψεων. Κάποιοι συνάδελφοι δεν ζήτησαν το λόγο. Κατ' εξαίρεση, μήπως να αρχίσω εγώ. Συμφωνείτε να κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων και μετά να απαντήσετε ομαδικά και σε λεπτομέρειες. Ωραία, μάλιστα. Μιλήσατε με ιδιαίτερο πάθος σε σχέση με την απελευθέρωση των θεωρήσεων και παρά τις ανησυχίες στα κρατημέλη μας είμαστε έτοιμοι να χορηγήσουμε στο κοσιοπέδιο ως τελευταία χώρα στην Ευρώπη απελευθέρωση των θεωρήσεων όμως ένας, μια προϋπόθεση είναι τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και θα ήθελα να γνωρίζω πότε η συνέλευση, η εθνοσέλευση του κοσυφοπεδίου θα ολοκληρώσει επιτέλους τις διαπραγματεύσεις. Πότε θα αποφασίσουν για τη συμφωνία περί συνόρων. Θα πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνουν πολλοί από εμά εδώ σε αυτήν την αίθουσα γιατί αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί από το κοινοβουλίο σας. Όταν ε, βλέπει κανείς τι θα πάρει ως αντάλλαγμα και είπατε ότι μάλλον είναι και το πιο σημαντικό θέμα της πολιτικής του, στην πολιτική ζωή του Κωσυφοπεδίου αυτή τη φάση. Ε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί τόσο αργείται. Ε, αυτό ζημιώνει και την εικόνα της χώρας. Πότε επιτέλους λοιπόν θα αποφασίσετε, φαντάζομαι, ε, από ό,τι κατάλαβα σήμερα πάλι συζητιέται στο Κοινοβούλιο, ίσως μπορείτε να μας πείτε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Και δεύτερη μου παρατήρηση. Εμείς όλοι εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την σημασία της συμφωνία των Βρυξελών που υπογράφηκε πριν από πέντε χρόνια. Εσεί το αναφέρατε σύντομα. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας ε, μιλά για τη δημιουργία μιας ένωσης κοινοτήτων ή ε, ε, δήμων στο Κωσυφοπαίδιο. Όμως δεν έχει υπάρξει ε, αρκετή πρόοδος σε αυτές τις σε αυτή τη διαδικασία με το Βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Πού βρίσκεστε λοιπόν και τι μπορεί, να τι μπορεί να κάνει η Πριστίνα ώστε να προχωρήσει το πράγμα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους δύο ειδικού μας για το Κωσυφοπαίδιο. Πρώτα τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας Ντανίνο Πίτσουλα. Ε, ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, καθώς ήρθατε και πάλι εδώ, δύο μήνες πέρασαν από τότε που συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο για την τέταρτη συνάντηση της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωσυφοπεδίου για τη σταθεροποίηση. Όπως θυμάστε τότε κάναμε μια εσβάθος και καρποφόρα συζήτηση για πολλά σημαντικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και ε, Σύνδεσης καθώς ε, και συζητήσαμε για την οικονομία, για την ε, καθορισμό των συνόρων με το Μαυροβούνιο, για τα εγκλήματα πολέμου, για το δρόμο προς την συμφιλίωση, της θεμελιώδης ε, ελευθερίας, την καταπολέμηση της οικιακής βίας, και επίσης σημειώσαμε από κοινού ότι φέτος το 2018 θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο παράθυρο ευκαιρίας για, την Ευρω... για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια και το Κωσυφοπαίδιο πιο συγκεκριμένα. Όμως δυστυχώς για πρώτη φορά δεν ε, καταλήξαμε σε κοινή δήλωση ή συστάσεις λόγω της έλλειψης συμφωνίας για το θέμα των ειδικών ε, ε, θεμάτων ε, επιμελητηρίων ε, και λόγω του ότι δεν υπήρξε τέτοια συμφωνία πιστεύετε πως θα έχει λυθεί το θέμα ε, μέχρι την δεύτερη ετήσια μας συνάντηση που θα γίνει στο Κωσυφοπαίδιο στο δεύτερο ήμιση του 2018. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η για το Κωσυφοπαίδιο, συνάδελφος Ίγκο Σόλτες που είναι από τους Πράσινους αλλά και είναι από την Σλοβανία. Σλοβενία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εξοχότατε. Πολύ αξιμών. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον καθαρισμό των συνόρων με το Μαυροβούνιο και την καταπολέμηση του διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος ε, και ούτω καθεξής. Πραγματικά θα θέλαμε να ακούσουμε από τη δική σας πλευρά αν μπορείτε να προβλέψετε αυτή την απόφαση που πραγματικά θα ανοίξει το παράθυρο ευκαιρίας για τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου, αλλά επίσης πρέπει να μας αναφέρουμε ότι είναι ένας από τους όρους που πρέπει να ε, τηρηθούν. Ο δεύτερος είναι η καταπολέμηση διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό που μας απασχολεί είναι τα σύνορα γιατί περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Πραγματικά πρέπει να σκεφτείτε τι παίρνετε ως αντάλλαγμα για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας περί συνόρων. Περιμένουμε με ανυπομονησία τη συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε και τις σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον. Και όπω είπε και ο κύριο Πίτσουλα, και εγώ θέλω να ρωτήσω Ποια είναι η κατάσταση προόδου. Ποια είναι η επίσημη θέση των αρχών του Κωσυφοπεδίου, ειδικά για αυτό το ειδικό επιμελητήριο. Ξέρουμε ότι η συζήτηση αυτή έχει μετακινηθεί στην Χάγη. Αλλά θα πρέπει να γίνει και παλήθευση των περιστάσεων του παρελθόντος, αλλά και μια νέα αντίληψη περί κράτους δικαίου και δημοκρατίας που είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουν οι επίσημοι φορείς και οι υποστηριχτές να στηρίξουν αυτό το ειδικό δικαστήριο για το κοσυφοπαίδιο. Είναι κρίσιμη η φάση για το κοσυφοπαίδιο. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι επίσης σημαντική. Ε, για να δούμε και πώς στην πράξη θα προχωρήσει η διαδικασία της απελευθέρωσης των θεωρήσεων ε, λοιπόν, ένα το θέμα είναι λοιπόν, είπαμε, τα σύνορα και μετά ε, τι θα γίνει με τα ειδικά δικαστήρια ε, του Κωσυφοπαιδίου. Ευχαριστώ πολύ. Πέτερ, Λεκούκον και Κουτσούκ είναι οι επόμενοι τρεις ομιλητές. Σωστά. Μάλιστα. Αυτοί οι τρεις ομιλητές λοιπόν και μετά θα δώσουμε το λόγο στον Υπουργό Εξωτερικών. Αλόης Πέτερλε από τη Σλοβενία, μέλος του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την ε, παρουσίασή σας. Πέρασε αρκετό διάστημα στο Κωσυφοπαίδιο τελευταία και με χαροποίησε η έμφαση που δώσατε στην πτυχή της σταθερότητας για το μέλλον. αλλά πιστεύω ότι η εσωτερική σταθερότητα του Κωσυφοπεδίου είναι σημαντική για τη σταθερότητα και ολόκληρη της περιοχής. Και βεβαίως θεωρώ πως αυτό το θέμα σχετίζεται πάρα πολύ με το, με το διάλογο με τη Σερβία. Εξού και η ερώτησή μου, τι ή ποια δυναμική μπορείτε να προβλέψετε Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου στηρίζεται από τη Σέρψκα λίστα επίση. Θυμάμαι τι συνέβαινε όταν η Σλοβενία προχωρούσε και διαπραγματευόταν την ένταξή της στην Ένωση, όπου ανταγωνιζόμασταν με τον εαυτό μας στην ουσία και νομίζω πως και το Κωσυφοπαίδιο είναι στην ίδια θέση, όπως και όλες οι άλλες χώρε χώρες υποψήφιες. Θεωρώ πως η ταχύτητα εξαρτάται πολύ από την ταχύτητα και την ποιότητα του διαλόγου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα περί αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Λόις Πέτερλε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Κιουτσούκ που τον γνωρίζετε νομίζω από τη, ε, σε και είναι από τη Βουλγαρία. Ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ, αγαπητοί συνάδελφοι. Και αγαπητέ συνάδελφοι, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκ μέρου τη ομάδα ALDE. Σα καλωσορίζουμε εδώ και χαιρόμαστε που σα βλέπουμε τόσο ενθουσιασμένο και για το Κωσυφόπεδο και για την Ευρώπη. Δεν θα καλύψω τα ίδια ζητήματα. Θέλω να κάνω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει. Ποια είναι η άποψή σα για την οικονομία, διότι είστε ένα από του πλέον γνωστού και επιτυχημένου επιχειρηματίε του Κωσυφοπεδίου και τη περιοχή. Κάτι που δεν συμβαίνει για γενικότερα όλους τους πολιτικούς στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω στοιχείο αυτό. Και δεύτερον, τι νέο φέρατε στη διπλωματία του Κωσυφοπεδίου από τότε που διοριστήκατε. Κατά την άποψή μου, το Κωσυφοπέδιο είναι μια σημαντική χώρα Ε, ε, έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Έχει τον νεότερο πληθυσμό στην Ευρώπη και θα πρέπει να συνεργαστούμε ολοκληρωμένα ε, με το Κωσυφοπαίδιο όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τέλος δίνω το λόγο στον Εντουαρτ Κούκαν από τη Σλοβακία επίσης μέλος της ομάδας του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριε Πρώτη Αντιπρόεδρε. Η χώρα μου, η Σλοβακία, δεν αναγνωρίζει επίσημα την ανεξαρτησία του Κωσυφοπηδίου, αλλά εγώ είμαι φίλος του Κωσυφοπηδίου και δεν χρειάζεται να σας δώσω άλλες εξηγήσει. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα, σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο αλλά να συνεργαστείτε και με τις πέντε μη αναγνωρισμένες χώρες, που δεν σας αναγνωρίζουν, να συνεργαστείτε μαζί, μαζί τους αντί να τις επικρίνετε. Ε, εγώ ξέρω ότι έχουμε σωστέ ε, σχέσεις με το Κωσυφοπέδιο, έχουμε ανταλλάξει κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείες και θεωρούμε ότι το μέλλον του Κωσυφοπεδίου είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Όλα τα άλλα σημαντικά ερωτήματα τέθηκαν ήδη από τους συναδέλφους μου. Όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, να πω απλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε ενεργά την απελευθέρωση, την απαλλαγή από θεωρήσεις. Είναι ένα θέμα που αφορά τους ανθρώπους, τα ανθρώπινα όντα και όχι θεσμικά όργανα. Και εδώ έχετε πέσει θύμα σαφώς διακριτικής μεταχείρισης. Είναι γεγονός. Χαιρόμαστε λοιπόν που αυτό θα αλλάξει και τώρα σας εκλυπαρούμε, κάντε τις τελευταίες κινήσεις, τα τελευταία βήματα, γιατί ε, κρατάτε τα πράγματα, ε, ε, δεν βοηθά τα πράγματα να προχωρήσουν. Κάντε κάτι, έχετε την μπάλα στη δική σας πλευρά του γηπέδου. Όσον αφορά και την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, μου έκανε δυσάρεστη έκπληξη ότι ήταν αδύνατο να καταλήξουμε σε κοινέ συστάσεις. Ξέρετε στην ιστορία του κοινοβουλίου αυτού, με την Τουρκία πάντα δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνίε. δυο Δύο-τρει φορές συνέβη με την Αλβανία και τώρα το κοσφοπέδιο βρίσκεται στην ίδια κατηγορία. Δεν είναι πολύ καλό αυτό. Και το ζήτημα μάλιστα που συζητούσαμε εκείνη τη στιγμή για το οποίο δεν καταφέραμε να επιτύχουμε συμφωνία είναι σημαντικό είναι σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα. Όσο το συντομότερο επιληφθεί θετικά και επικοδομητικά από πλευρά σας, τόσο το προτιμότερο. Τόσο το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ασχοληθήκατε με όλα τα ζητήματα. Ήσασταν πολύ πλήρης. Ξέρουμε όλοι ότι το Κοσφοπέδιο έχει το νεότερο λαό της Ευρώπης. Πολύ δυναμικό. Και είμαι βέβαιος ότι τους αξίζει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό μέλλον. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να σας δώσουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη, αλλά και εσείς θα πρέπει να βοηθήσετε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Thank you, Edward Kukan. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Edward Kukan. Δεν υπάρχουν άλλοι μιλητές στο κατάλογο, οπότε... Κύριε Αντιπρόεδρε, όπως είπαν οι συναδέλφοι, τα βασικότερα ζητήματα που έχουμε στην Επιτροπή αυτή με τη χώρα σας είναι το σύνορα με το Μαυροβούνιο, το ότι θέλουμε να συνεχίσετε την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και οι εργασίες του ειδικού σώματος ε, για την απονομή δικαιοσύνη. Θα ήθελα να κάνω και άλλες δύο ερωτήσεις, πριν αυτό που έκανα στην αρχή. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τα εξή παρατηρείται καθόλου πρόοδος για τη δολοφονία του κυρίου Ιβάνοβιτς. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Και τέλος, αναφέρατε αναφέρατε ότι είναι χαμηλός ο αριθμός των ετούντων άσυλο, έχει μειωθεί 7.000. Μιλάμε για ανθρώπους που κινούνται προς τη Βόρεια Ευρώπη, ε, προς τη χώρα προς τη Γερμανία. Μειώστε τον αριθμό από 70.000 στις 7.000. Αλλά η ερώτησή μου είναι γιατί υπάρχουν ετούντες άσυλο από το κοσυφοπαίδιο. Η χώρα σας είναι μια ελεύθερη χώρα, είναι μια δημοκρατία, είναι μια ασφαλής χώρα καταγωγής. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι ετούνται άσυλο. Γιατί εξακολουθούν να ετούνται άσυλο στην Ευρώπη. Ποια είναι η στάση σας γι' αυτό και τι κάνει η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου ώστε να ενθαρρύνει τους πολίτες του Κωσυφοπεδίου να μην προσπαθούν καν να κάνουν αίτηση ασύλου σε χώρες όπως η Γερμανία, διότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να γίνουν δεκτές οι αιτήσει τους. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που είχαμε να σας κάνουμε. Έχετε το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, κύριε Κούκα, μου δώσατε λίγο θετική ενέργεια. Ε, τη χρειαζόμουν σήμερα. Ευχαριστώ. Και κύριε Μακάλιστερ, λοιπόν, θα ξεκινήσω από την υπόθεση Ιβάνοβιτς, ο οποίος ήταν φίλος μου. Τον γνώριζα από το 2005. Έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές, συναντηθεί, και συμφάγει. Γνώριζα την οικογένειά του και λυπάμαι απεριόριστα που δεν τον έχουμε πλέον μαζί μας. Την ημέρα της δολοφονίας του θυμήθηκα τι μου είχε πει παλιότερα. Μου είχε πει ότι κάποια μέρα κάποιος θα με σκοτώσει. ήταν μια έμονη ιδέα του ότι κάποια στιγμή κάποιος θα τον δολοφονήσει. Και όταν του λέγαμε μα είναι δυνατόν ποιος θα σε σκοτώσει έλεγε η Σέρβη μου έλεγε και πιστεύω ότι είχε δίκιο σίγουρα δεν τον σκότωσαν Αλβανοί και ελπίζω πολύ πολύ σύντομα να έχουμε στα χέρια μας το όνομα του δολοφόνου. Και θα δούμε ότι δεν ήταν ε, λόγω σύγκρουσης μεταξύ εθνοτήτων. Γιατί, γιατί ο τη της Μητρόβιτσα σήμερα είναι όπως στη δεκαετία του 80. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουμε καμία πρόσβαση ή ελάχιστη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εκεί για αυτό το κομμάτι του κοσφοπεδίου. Πρέπει να απελευθερωθεί όμως. Και όταν εννοώ να απελευθερωθεί εννοώ από εγκληματίες και των δύο πλευρών πιθανότητα, όχι μόνο Σέρβων και Σέρβων και Αλβανών, ε, οι οποίοι είναι εγκληματίες. Όταν εγώ ήμουν πρόεδρος την τρίτη μέρα πήγα στο βορρά και ήμουν ο πρώτος και πιθανότατα ο τελευταίος αξιωματούχος από το κοσυφοπαίδιο που πήγε στο βορρά. Και περπατούσα εκεί στους δρόμους και με σταματούσαν μεγάλες γυναίκες ηλικιωμένες και μου έλεγαν «Ο γιο μου σας παρακαλώ, γέ μου σα παρακαλώ, κάντε κάτι, υποφέρουμε από του εγκληματίε και από τις δύο πλευρέ και από του Αλβανού και από του Κοσοβάρου. και από από όλους. Ε, κοιτάξτε, μας κοιτάνε τώρα. Λυπάμαι τόσο πολύ για αυτό που συμβαίνει στο Βαρά. Λυπάμαι τόσο πολύ για τον Ιβάνοβιτς. Αλλά ελπίζω ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι θα έχ... βρούμε το όνομα, τα ονόματα των ανθρώπων που τον δολοφόνησαν. Όσον αφορά τους μετανάστες μας, τους μετανάστες από το Κωσυφοπέδιο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Όλοι πιστεύω γνωρίζουν ότι το Κωσυφοπαίδιο είναι μια δημοκρατική χώρα. Δεν υπάρχει πολιτική πίεση πουθενά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φύγει κανείς από το Κωσυφοπαίδιο. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι η οικονομία. Είμαστε, βλέπετε, μια χώρα που ήμασταν ανοιχτοί ε, τα δεκαετία του 70, του 80, στην αρχή της δεκαετίας του 90 οι άνθρωποι είναι πολύ λέει. πολύ δραστήριοι, θέλουν να προοδεύσουν, να δημιουργήσουν ένα μέλλον και τώρα είναι αποκλεισμένοι. Είναι σαν μια μαύρη τρύπα των Βαλκανίων. Και πιστεύω, ξέρετε, όταν κηρύξαμε την ανεξαρτησία μας το 2008 από τότε, δεν υπήρξε άλλη σύραξη μεταξύ εθνοτήτων στο κοσυφοπαίδιο. Την ημέρα λοιπόν που θα υπάρξει η απαλλαγή από τις θεωρήσεις είμαι βέβαιος ότι κανένας δεν θα ξανάρθει να ζητήσει άσυλο εδώ. Αυτό είναι βέβαιο. Διότι θα το είδατε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι ήρθαν πίσω. Είχαν τη δυνατότητα να πάνε στη Δύση, αλλά ήρθαν πίσω. Έτσι είναι η νοοτροπία στη χώρα μας και πιστεύω ότι τη στιγμή που θα υπάρξει απαλλαγή από θεωρήσεις για το κοσυφοπαίδιο, οι κάτοικοι του κοσυφοπαιδίου θα πάψουν να αναζητούν, να επιδιώκουν να, λάβουν άσυλο. Θα πάψουν να υπάρχουν αιτούντες άσυλο. Τώρα για τα σύνορα. Η οριοθέτηση αυτή χρειάζεται να παρέσει από το Κοινοβούλιο να ακυρωθεί. Όχι σήμερα, εχθέ, έπρεπε να έχει γίνει πριν από τρία χρόνια. Γιατί, διότι έχουμε ένα περίεργο συνδυασμό δυνάμεων στο Κοινοβούλιο. Η αντιπολίτευση ανέκαθεν ήταν 50%. Και είχαμε κιόλας βουλευτές που δεν ήταν απολύτως αβέβαιοι για το κατά πόσο θα ψηφίσουν. Η οριοθέτηση αυτή το σύνορο υπήρχε μια ευκαιρία να ψηφιστεί το 2015, αλλά χάθηκε η ευκαιρία και σήμερα αντιμετωπίζουμε σοβαρότατε δυσκολίε γιατί χρειαζόμαστε δύο τρίτα των ψήφων των βουλευτών. Ήταν αδύνατο να επιτευχθεί τέτοια πλειοψηφία ακόμη και σήμερα. Το τελευταίο τρίμηνο εργαζόμαστε σκληρά για το θέμα αυτό. Πριν από 10 μέρες κατέστησα φες ότι η κύρωση θα λάμβανε χώρα. Γιατί είχαμε λάβει σχετικές ε, υποσχέσεις από το Ριστασέφικα, αλλά τελευταία στιγμή αποσύρθηκαν. Διότι βρίσκονται υπό την ισχυρή επιρροή του Βελιγραδίου. Πιστεύω, εγώ, μπορεί και να μην έχω δίκιο, αλλά δεν είναι οι μόνοι που μπλοκάρουν το σχέδιο. Ναι, φυσικά. Έχουμε και τους δικούς μας ε, εξτρεμιστές που δεν πρόκειται ποτέ να υπερψηφίσουν αυτή τη συμφωνία. Αλλά και η αντιπολίτευση ε, δεν πρόκειται ποτέ να λάβει την εξουσία στο κοσικό πεδίο γιατί ο κόσμος δεν τους θέλει. Το... Σήμερα έχουν το μέγιστο που μπορούν να επιτύχουν από ψήφου και έχουν χωριστεί και στα δύο. Οπότε ελπίζουμε αυτό το μετριοπαθέ κομμάτι να υποστηρίξει το πέδιο στα σημαντικά ζητήματα. Και εγώ είμαι έτοιμο, ελπίζω σήμερα ότι στι 4 η ώρα θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σήμερα στι 4. Ναι, το κοινοβούλιο μας. Ελπίζουμε, ελπίζω είπα, Ελπίζω ότι θα ευοδοθεί ψηφοφορία. Θα δούμε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι μία από αυτές τις ημέρες θα, θα κυρωθεί η οριοθέτηση το, τα σύνορα. Ε, τώρα μια ερώτηση του κυρίου Πίτσουλα αφορούσε το ειδικό δικαστήριο. Ναι δεν ήταν ωραίο. Ήταν μια άσκημη έκπληξη, διότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από τους, ε, από τους βετεράνους. Αυτοί παρουσίασαν την πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο έλαβαν μεγάλη υποστήριξη. Ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο. Εκείνη την εποχή εγώ ήμουν ε, σε ταξίδι στην Αφρική και Μόλις ε, έλαβα την πληροφορία, ζήτησα από τους βουλευτές μου, του υπουργού μου, να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση. Τελικά επιλύσαμε το πρόβλημα με μεγάλη πίεση από τη Δύση, από τις Βρυξέλλες, από τη ΣΥΠΑ και σήμερα μπορώ να σας πω ότι το πρόβλημα αυτό έχει λήξει. Ή μάλλον έχει περάσει, δεν έχει τελειώσει ολοκληρωτικά, αλλά πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει ε, στι ε, συζητήσεις μας. Έχει λήξει πιστεύω το πρόβλημα του δικαστηρίου αυτού. Αλλά όλα τα μέρη πρέπει να αρχίσουν να κάνουν κάτι, γιατί το έχουμε συζητήσει τόσο πολύ αυτό το ειδικό δικαστήριο, ε, σχεδόν τέσσερα χρόνια. Τόσο που κανείς δεν, και ξέρετε, κανείς δεν το εμπιστεύεται. δεν έχουν κάνει και τίποτα. αν θέλουν να κάνουν. Ε, ξέρετε, πρέπει να πούν αφού ότι δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία, ούτε πρόκειται να βρουν για όλα αυτά που ισχυρίζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί βρισκόμαστε. Εδώ βρισκόμαστε. Το ζήτημα είναι λήξαν. Κυρίε κύριοι, ε, μιλήσετε για τα σύνορα. Ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Εγώ έχω, σας έχω στείλει τόσες πολλές φορές πληροφορίες για την κατάσταση. Και την τελευταία φορά που σας έκανα ενημέρωση ήμασταν πολύ κοντά. Είχαμε το OK από τη λίστα σας και τη λίστα και τελικά θέτησαν την υποσχέσή τους. Ελπίζω λοιπόν ότι σήμερα θα τα καταφέρουμε. Ελπίζουμε σήμερα ότι θα είναι η ευτυχή σήμερα που θα λήξει το ζήτημα για το ειδικό δικαστήριο. Επίσης είμαι βέβαιος ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί άλλο με αυτό το ζήτημα. Το ειδικό δικαστήριο λοιπόν θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Uh, Κύριε Πέτερλε, γνωρίζετε πολύ καλά πώς έχει κατάσταση όταν γίνεται λόγος για την ανεξαρτησία του Κωσόβου. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι και το σύνταγμά μας είναι πάρα πολύ περίπλοκο και ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε δύο τρίτα ε, πλειοψηφία μόνοι μας, χωρίς τους Σέρβους. Οι οποίοι Σέρβοι λένε όχι σε όλα ουσιαστικά όταν έρχονται στη Βουλή για, ή ε, στη δημιουργία των θεσμών στην οικοδόμηση του κράτους για σημαντικά θέματα. Διάλογος Πρίστινας Βελιγραδίου. Uh, Έχουμε διάλογο με τους Σέρβους. Ο πρόεδρός μας προετοιμάζει το επόμενο βήμα. Υπάρχει χρονικός περιορισμός. 20 χρόνια το συζητάμε με τους Σέρβους περίπου. Αυτή τη φορά μάλλον θα πρέπει να βάλουμε κάποιο χρονικό όριο με πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα να συζητήσουμε με τους Σέρβους. Ξέρετε, αυτά που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες, γιατί είναι πολλά τα εμπόδια στην καθημερινή μας συμβίωση με Σερβία. Αλλά αυτός ο διάλογος θα πρέπει να λάβει υπόψη του δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει το Κωσοβό σε ανεξάρτητο κράτος και ουδής μπορεί να το παραγνωρίσει αυτό ή να το αγνοεί. Και το δεύτερο γεγονός είναι ότι η Σερβία είναι παράγον σταθερότητα στο βόρειο Κωσυβοπαίδιο και όλοι πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουν και να το αποδεχθούν. Κινώντας λοιπόν από αυτά τα δύο δεδομένα θα πρέπει εμείς να χτίσουμε το μέλλον μας όπου είναι μια συμβίωση με τους Σέρβους. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν μπορούμε να βάλουμε σύνορα μεταξύ των δύο αυτών πληθυσμών. Είναι μεικτοί οι πληθυσμοί. Πολλοί Σέρβοι ζουν στο Κόσοβο και έχουν ε, οικογένειες στη Σερβία. Και Τούμπαλεν. Και πολλοί Αλβανοί που ζουν ε, στη Σερβία έχουν οικογένειες στο Κόσοβο. Δεν μπορούμε κάθε μέρα. Ε, αυτοί οι άνθρωποι περνούν τα σύνορα καθημερινά. Και θα πρέπει να εγγυηθούμε αυτή τη συμβίωση στους λαούς μας και να επενδύσουμε στην οικονομία. Αυτό είναι το βασικό. Δεν μπορούμε απλώ να λέμε στου Σέρβου δεχτείτε την ανεξαρτησία του Κωσόβου. δεν πρόκειται ποτέ να τη δεχτούν. Εάν όμω έχουμε κάτι να του προσφέρουμε, τότε μπορεί και να το σκεφτούν. Γιατί στο βόρειο Κόσοβο Έτσι όπως έχει η κατάσταση δεν μπορούμε να πετύχουμε ποτέ τίποτα. Θα πρέπει η οικονομία να κινηθεί. Και εγώ πάντα πίστευα ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ζώνη ελευθερών συναλλαγών μεταξύ Σερβίας και πεδίου. Το Σάββατο συναντήθηκα με τον κύριο Τάτσης, ε, τον Ήβιτσα Τάτσης, ναι, και το συζητήσαμε στο Σαράγεβο. ας πούμε σε χονδρικά να δούμε την Νότια Σερβία και το Βόρειο Κωσυβοπέδιο και να δημιουργήσουμε μια ελεύθερη οικονομική ζώνη για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση εκεί. Και πραγματικά σίγουρα θα αλλάξει. Γιατί σε τελική ανάλυση τι χρειάζεται ο κόσμος καθημερινά ασφάλεια, μεγαλύτερο εισόδημα, καλύτερη ζωή και τίποτα παραπάνω. Και πραγματικά ο κόσμος στο βορρά του Κωσόβου χρειάζεται ασφάλεια, καλύτερα σχολιά, ε, περισσότερα εισοδήματα και καλύτερο ποιοτικό επίπεδο. Για αυτή την οικονομική ζώνη λοιπόν ελευθερών συναλλαγών το συζήτησα με τον κύριο Ντάτσιτς Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δοθεί συνέχεια, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες εκεί. The ε, χωρίς να φύγει η ε, κυριαρχία των δύο χωρών, μπορούμε να οικοδομήσουμε κάτι πραγματικά χρήσιμο και εφικτό. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί φέτος, μέχρι τα τέλη του έτους, για να έχουμε ένα ειρηνευτικό σύμφωνο ε, με τη Σερβία. όπου να αναγνωρίζει η Σερβία το γεγονός ότι το Κόσοβο υπάρχει ως ανεξάρτητη χώρα δεν μπορεί να το παραγνωρίζει, να το αγνοεί και το Κόσοβο θα πρέπει να αναγνωρίσει επίσης ότι υπάρχει η Σερβία. Και είναι πολύ σημαντικός εταίρος για μας. Ο κύριος Κιουτσούκ αναφέρθηκε στην οικονομία. Όταν ανέλαβα στην κυβέρνηση, είχα μεγάλο ενθουσιασμό και ικανοποίηση ότι θα επιτύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά τώρα έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες και έχει αποσπαστεί κάπως η προσοχή μας από τις μεταρρυθμίσεις που επιβραδύνθηκαν. Πάντως σίγουρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις στο κοσυφοπαίδιο. Χρειάζεται μια οικονομία που να αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύς πάνω από 8%. Αν αναπτυσσόμαστε με ρυθμούς κάτω του 8% δεν κάνουμε τίποτα για τον κόσμο, απλώς αλλάζουμε συνάλλαγμα. Δηλαδή λεφτά που αλλάζουν χέρια, δεν κάνουμε τίποτα για τον κόσμο. Χρειαζόμαστε ελεύθερες οικονομικές ζώνες για να λειτουργήσουμε αλλά και γεωργία. Η γεωργία είναι μεγάλη ευκαιρία για το Κόσοβο. Αλλά στη γεωργία χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια. Ένα είδος ε, σχέδιο Μάρσαλ. Εργαζόμαστε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και στο συγκεκριμένο πεδίο. Μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Βεβαίως. Πολλά αλλάζουμε. Πολλούς πρέσβες μεταθέτουμε. Ναι, ο Μπέρναρτ. Εσύ επέζησες, πάλι καλά. Ωραία, ευχαριστή είδηση λέει ο πρέσβης. Αλλά στο εσωτερικό των υπηρεσιών μας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάνουμε κάποιες ανακατατάξεις. Και έχουμε δώσει την εντολή στους πρέσβες και στους διπλωμάτες να μην απαντάμε σε προκλήσεις της Σερβίας να μην απαντάμε. Είδαμε ότι είναι καλύτερη τακτική αυτή. Άστο να πέσει κάτω παρά να απαντήσει στην πρόκληση. Και όποιος θέλει να έρθει στο κοσυφοπαίδιο μπορεί να έρθει ανα πάσα στιγμή και πολιτικοί να έρθουν όποτε θέλουν είμαστε πάντα πάρα πολύ ευγενείς απέναντί τους. Έχουμε και διάφορες πρωτοβουλίες στο Υπουργείο μας. Συστήσαμε μία επιτροπή για την προαγωγή και πρόθεση της ειρήνης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Καμία σχέση αυτό με το διάλογο. Αλλά για την προαγωγή της ειρήνης μαζί με τη Σερβία. Διοργανώνονται συναυλίες, συνεδριάσεις, εκδηλώσεις, σκηνές όπου συμμετέχουν διάφορες ομάδες ε, ενδιαφερομένων και συμφερόντων. Και πραγματικά έχουμε κάποια αποτελέσματα εκεί. Επίσης, έχουμε κάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό του Υπουργείου. Θα μπορώ να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Κωσοβού είναι πάρα πολύ δυναμικό, δραστήριο και ενεργό σήμερα. Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά όμως γι' αυτό. Κύριε Κούκαν, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τις εξηγήσεις σας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τις πέντε χώρες που δεν μας έχουν ακόμα αναγνωρίσει. Και ξέρουμε ότι έχουμε φίλους στις χώρες αυτές. Στη Σλοβακία, για παράδειγμα, η οποία ανέκαθεν ναι, μας υποστηρίζει, ήταν ευγενική μαζί μας. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Ε, πιστεύω ότι κάποια μέρα θα έρθει αυτή η μέρα που θα μπορέσουμε να προσβλέπουμε στη φιλία μας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Βλέπετε, κύριε Μακάλιστερ, ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και είμαστε και λίγοι αριθμητικά. Πάντως, αποβούληση είναι δεδομένη αυτή. Κύριε Υπουργέ Πατσόλη, εξ ονόματος των μελών της Επιτροπής μας, σας ευχαριστούμε που ήρθατε στις Βρυξέλλες ε, και εκτιμούμε την ειλικρίνειά σας, ώστε να σας χειροκροτήσουμε γιατί το αξίζετε. We are Προσβλέπουμε στις μελλοντικές μας συνεργασίες και, και επαφές και Ελπίζουμε να μάθουμε καλά νέα από την Πρίστινα ότι θα κυρωθεί η συμφωνία ε, για την ορθέτηση των συνόρων με το Κωσυφοπέδιο με το Μαυροβούνιο. Να έχει θετική έκβαση. Αυτό θα ήταν πολύ καλό και θα διευκόλυνε πάρα πολύ τα πράγματα. Και πάλι καλή σας μέρα στις Βρυξέλλες. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στην Επιτροπή μας κάποια στιγμή. Colleagues, we will continue our meeting in five minutes. Σε πέντε λεπτά συνεχίζουμε, συνάδελφοι. So, Κυρίες και κύριοι, επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι το υπαριθμό 16. Να καλωσορίσουμε θερμά τον δόκτωρα Ρενάτ Μανσούρ, ερευνητή στο Chatham House για θέματα Βόρειας Αφρικής. και έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης που ανατέθηκε από την Επιτροπή ΑΦΕΤ με θέμα ανοικοδόμηση του Ιρακινού κράτους, σταθεροποίηση, διακυβέρνηση και συμφιλίωση. Δόκτωρα Μασούρ, η μελέτη σας ε, ολοκληρώθηκε σε πολύ κατάλληλη στιγμή. Εμεί ασχολούμαστε με την ε, ολοκλήρωση της, συνεργα... της ε, συμφωνίας ε, συνεργασίας με το Ιράκ. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σαΐφη. Και βλέπουμε πως η συμφωνία αυτή είναι αβέβαιη ως προς το μέλλον της. Έχουμε επαφή με το Κουβέιτ και το Ιράν ενώ συγκαλούσαμε τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση του Ιράκ. Μάλιστα και στο ίδιο ξενοδοχείο γινόταν εκεί που μείναμε. Και μάλιστα τρακάραμε τον Επίτροπο του Στυλιανίδη προς έκπληξή μας. Λοιπόν, έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. 12 και 40 το αργότερο πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Εγώ θα περιοριστώ στα 10 λεπτά ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και ερωταπαντήσεις και να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση των ερωτήσεων, των απορριών που μπορεί να έχετε για... καθώς προχωράμε. Γιατί όπως είπε ο κύριος Μακάλιστερ υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας αυτή τη στιγμή στο Ιράκ ε, σε αυτό που ο κόσμος αποκαλεί μετα εποχή μετά ίσης, τα συγκρουσιακή εποχή. Εμείς βέβαια οι πανεπιστημιακοί αποφεύγουμε τέτοιου είδου ε, εκφράσεις γιατί το έχουμε δει και παλιότερα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στο Ιράκ είναι ότι ακριβώς έχουμε δει αυτούς τους κύκλους νοικοδόμησης ε, και μετά αποτυχίας. Οπότε το θέμα πρέπει να είναι πώς αποφεύγουμε τα ίδια λάθη. Αν δούμε το 2008-2009 θα είχαμε την ίδια ακριβώς συζήτηση, αλλά τότε ήταν η Αλκάιντα και το Ισλαμικό κράτος. Τώρα μιλάμε για την μετά Νταές εποχή. Πώς θα αποφύγουμε λοιπόν τα ίδια λάθη το περιοδικό Time σίγουρα έκανε λάθος όταν ε, είπε ότι τέλος το Ιράκ. Ε, σαφώς δεν τελείωσε η υπόθεση του Ιράκ, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι. Πριν από ένα μήνα γύρισα, πέρασα πολύ καιρό στην Παγδάτη, στο Μοσούλη, και τα λοιπά, προσπάθησα να καταλάβω τι συμβαίνει στο κέντρο, τι συμβαίνει στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Και στο έκθεση αυτή που συνέταξε το βασικό μου επιχείρημα είναι ότι νομίζω πως ο ρόλος της Ένωσης πρέπει να είναι να οικοδομηθούν θεσμοί και όχι προσωπικότητες. Πάντοτε θεωρούμε πως είναι δύσκολη η ε, σύσταση ενός κράτους ε, σε ολόκληρο τον κόσμο όπου η διεθνή κοινότητα πρέπει να κατασκευάσει στην ουσία ένα κράτος και θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στους θεσμούς και όχι στις προσωπικότητες. Αυτό σημαίνει η οικοδόμηση του κράτους. Όλα τα υπόλοιπα από αυτό εξαρτώνται. Έχουμε διάφορες λέξεις που ακούγονται διαρκώς από το 2003 Δηλαδή η συμπερίληψη, η inclusivity, τα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιούσαν συνέχεια αυτή τη, τη λέξη. Τι σημαίνει inclusivity, δηλαδή οι Σουνίτες, οι Ιτες, οι Χριστιανοί όλοι μαζί. Ναι, αλλά τελικά ε, φτιάχτηκε ένα σύστημα της ελίτ έναντι στου πολίτε που το αφισβητούν οι ίδιοι οι Ιρακινοί. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε με αυτό το είδος την ε, διαδικασία νομιμοποίηση από πάνω προς τα κάτω. Όταν μιλάμε για συμφιλίωση για παράδειγμα, μιλάμε για του Ιήτε και τους Σουνίτε μαζί, έναν ηγέτη, δύο ηγέτε μάλλον που θα πρέπει να κάτσουν δίπλα-δίπλα και να πούμε άρα ότι ναι, το Ιράκ μπήκε στο σωστό δρόμο. Γιατί τα μεγαλύτερα χάσματα το μεγαλύτερο χάσμα μάλλον που ισχύει είναι ανάμεσα στους πολίτες και στην ελίτ. Πραγματική συμφιλίωση σημαίνει λοιπόν ε, γεφύρωση αυτού του χάσματος. Δεν πρέπει δηλαδή να ενισχύονται οι ταυτότητε ενώ το Ιράκ προσπαθεί να κινηθεί. Από το 2015 έχουμε τους, ε, τους ε, στη Βασόρα που διαμαρτύρονται κατά των ε, ε, ηγετών τους και τους Σουνίτες που διαμαρτύρονται κατά των δικών τους ηγετών. Δηλαδή δεν μπορούμε να βασιστούμε στα όσα ξέραμε παλιά προσπαθώντας να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Για να μην φτάσουμε σε ένα νταές ε, νούμερο 2. Ε, πρέπει να συνδυάσουμε δηλαδή το, το επίσης το βραχυπρόθεσμα με το μακροπρόθεσμα πολιτική. Αν δούμε ας την πολιτική την αμερικανική σε σύγκριση με την ιρανική πολιτική στο Ιράκ θα δείτε τεράστια διαφορά ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες σκέψεις της Αμερικής α, ε, που επηρεάζονται κάθε φορά από τις επόμενες εκλογές ενώ το Ιράν κοιτάει τι θα γίνει σε 10-20 χρόνια και να προσπαθήσουμε αυτά να τα συνδυάσουμε. Άρα λοιπόν εγώ στην μελέτη μου τα εξετάζω και τα δύο και, προσπαθώ να δω πώς μπορούμε αυτό να τα συνδυάσουμε. Εγώ επέστρεψα μόλις από τη Μοσούλη. Η κατάσταση της ασφάλειας είναι καλή για την ώρα, αλλά μπορεί κανείς να δει ότι κανείς δεν ξέρει που είναι το γενικό επιτελείο. Υπάρχουν ένα σωρό καταστάσεις που μας κάνουν να διερωτηθούμε για το πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση της ασφάλειας. Τώρα, σε άλλα μέρη του Ιράκ, ε, μπορεί να δεις την, ότι αναδύεται και πάλι το, το ISIS, ε, όπως το Κυρκούκ, ας πούμε. Δεν θέλουμε λοιπόν να τους βομβαρδίσουμε ε, απαραίτητος, αλλά πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά. Τώρα, οι υπηρεσίες σε πολλές περιοχές. Αυτό που είναι σημαντικό για τον πολίτη δεν είναι ε, να συναντηθούν ε, οι ηγέτες μεταξύ τους, αλλά το να έχουν ηλεκτρισμό, νερό, υπηρεσίες, ένα κράτος σε βάση περιπτώσει που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και να τους εκπροσωπεί. Ε, αυτά είναι τα θέματα τα πιο σημαντικά. Δηλαδή να έχεις ένα θεσμό που πιστεύεις ότι σε αντιπροσωπεύει, ότι δηλαδή ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες και ε, τώρα, αν μιλήσουμε για την, τον, τον, την επιστροφή των εκτοπισμένων, οι περισσότεροι με τους οποίους εμείς συνομιλούμε, οι συζητήσεις μιλάνε για δουλειά, για χρήματα, για αποκατάσταση των ζωών τους. Αυτές είναι, η είναι η για την ανοικοδόμηση του κράτους. Αυτές είναι πιο βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Οι πιο μακροπρόθεσμε είναι πιο περίπλοκέ, αλλά πάρα πολύ σημαντικέ, γιατί οι βραχυπρόθεσμες μας δίνουν ε, μικρές και σύντομε νίκες, ενώ μακροπρόθεσμα θα έπρεπε να είναι, πιο δύσκολο. Σήμερα εορτάζεται η 15η επέτειος της εισβολή στο Ιράκ. Αν είχες πει στου ε, πολίτες της Ένωσης ε, ή τη Αμερική ότι ότι αν πας αυτό το πόλεμο μέχρι το 2018 εκεί θα είσαι, οι περισσότεροι θα λέγανε όχι, λάθος κάνετε. Άρα λοιπόν αυτή είναι η τραγωδία, ότι δεν είδε κανείς το μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τώρα, κάποιο πολύ σημαντικά θέμα είναι η διάχυση της εξουσίας. Άλλος ένα, άλλη μια λέξη που ακούγεται συνέχεια, η αποκέντρωση. Η ιδέα για μετά το 2003 ήταν ότι οι τοπικέ κυβερνήσει ε, και οι τοπικέ αρχέ θα μπορούσαν να τοποκριθούν καλύτερα στι ανάγκε των πολιτών από την κεντρική, τρα... Ε, κεντρική διοίκηση. Γιατί οι περισσότεροι ε, που ανοικοδόμησαν, είτε οι Σιήτε είτε οι Κούρδοι, είχαν πραγματικά τραυματικέ εμπειρίε για το τι σημαίνει κεντρικό κράτο και προσπάθησαν να φτιάξουν ένα αδύναμο κράτο, ώστε οι εξουσίε να είναι αποκεντρωμένε. Ε, γι' αυτό μπορούσε να χαθεί εξουσία και να αναλυφθεί από ομάδες όπως το ίσις ε, και αυτό βλέπουμε από την ιστορία μετά το 2013. Ε, Άρα λοιπόν είναι πιο αντιπροσωπευτικό να έχουμε τοπικές αρχές. Πώς μπορεί μια κεντρική κυβέρνηση ω θεσμό να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες από την Βασόρα μέχρι τη Μοσούλη, μέχρι τη Σουλεϊμανία. οι Κούρδοι ας πούμε, χρησιμοποιούν ε, περισσότερο τη φράση ομοσπονδιακή κυβέρνηση αντί για κεντρική κυβέρνηση. Ε, Ακριβώ λόγω αυτών των ταμπού και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Μεταρρύθμιση τώρα του τομέα τη ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Ιράκ, ειδικά ε, στις περιφέρειες, υπάρχουν διάφορες ένοπλε δυνάμει που προέκυψαν πριν ε, αλλά και μετά από το ΆΣΙΣ 2. Ε, αυτοί εδραιώνονται νομικά, πολιτικά, οικονομικά έχουν ε, ε, δημιουργηθεί διάφορες ομάδες και αποτελούν κομμάτι του κράτους. Το θέμα δεν είναι ότι αυτές οι ομάδες θέλουν να είναι μέρη του ίδιου του κράτους, αλλά ότι υπάρχουν φορείς που μπορούν να κινούνται σε μια φαιά ζώνη και διαλέγουν πότε θα είναι μέσα στο κράτος και πότε θα είναι παρακρατικοί. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός λοιπόν τι είναι κράτος και τι όχι και άρα αυτοί παίζουν σε διάφορα ταμπλό. Όταν ανέλαβε ο Μαλίκη, πήγε στο γραφείο του και πήρε το, το CTS μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Αλλά υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις, γι' αυτό γιατί λέγανε ότι ήταν αντισυνταγματικό. Όμως τώρα λένε ότι αυτό το κομμάτι είναι κρατικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο Κοινοβούλιο, γιατί εκεί ε, γίνεται η νομοθεσία. Δυστυχώ στο Ιράκ υπάρχουν δύο εμπειρίε από το κοινοβούλιο. Έχουμε το κοινοβούλιο του Κουρδιστάν που δεν ε, συνεδρίασε για δύο χρόνια ή το Ιρακινό κοινοβούλιο όπου οι πολιτικοποίηση συμφερόντων και τα λοιπά μπόρεσαν να προωθήσουν τι δικέ τους ατζέντε. και πάλι αυτό επανέρχεται στην εκλογική μεταρρύθμιση. Πώς φτάνει κανείς στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο εστιάζουν οι Ρακινοί. Δεν έχει γίνει ακόμα. Για τις επόμενες εκλογές όμως πρέπει να γίνει η εκλογική μεταρρύθμιση. Και όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να σας μιλήσω για όλα αυτά σε 10 λεπτά, αλλά φαντάζομαι ότι στην σύνοψη θα δείτε ότι πιστεύω πως αυτό που πρέπει να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τις παγίδες της οικοδόμησης κράτους από πάνω προς τα κάτω είναι να είμαστε πιο ε, δραστήριοι και πιο ε, αργή γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε στις μακροπρόθεσμες ανάγκες περισσότερο. Το να ανταποκρινόμαστε ε, ανα πάσα στιγμή στις πρόσκαιρες απαιτήσει δεν ωφελεί. Και επίσης ε, να, με το μαλακό να προχωράμε. Thank you. Εγώ ευχαριστώ κύριε Μανσούρ. Γιατί σύντομη κατά τα άλλα παρουσίασή σας. Ανταλλαγή απόψεων τώρα. βεβαίω, θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Τσαϊφή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μασούρ, ιδιαίτερα για την παρουσία του εδώ, αλλά και την ποιότητα της έκθεσης ε, και της μελέτης. Ε, το Δεκέμβριο του 2017 κρυζώθηκε από την επικράτεια εκεί ο Άισις και τώρα το 2018 θα πρέπει να είναι το έτος ανοικοδόμησης ενός ασφαλού, σίγουρου και συμφιλειωμένου κράτους. Οι στόχοι της ασφάλειας, ε, της συμφιλίωσης ε, και της ανοικοδόμησης της ε, χώρας είναι αλληλένδετοι και θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν. Η σταθεροποίηση της χώρας δεν μπορεί να γίνει παρά ε, μόνο μέσα από την αδιάρθρωση της αστυνομίας. Θα πρέπει να επανέλθουν οι υπηρεσίες πρώτης ανάγκης και να είναι σίγουρη και αντιπροσωπευτική η διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο και εθνικό χωρίς αποκλεισμούς. Είναι πολλές οι προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό Δημοσίευση και έγκριση κοινή στρατηγική για το Ιράκ και δέσμευση όλων των θεσμικών οργάνων είναι δεδομένη. Ε, ε, στο Κουβέιτ το Φεβρουάριο εκφράστηκε αυτό και τώρα θα πρέπει να μεταφραστεί στην πράξη ε, με δράση υπέρ χώρα. Είναι επίγον να επανέλθουν οι υποδομές, να γυρίσουν σε στήρε εσωτερικά εντοπισμένοι, εκτοπισμένοι σε χώρες και χώρους που απελευθερώθηκαν πρόσφατα ε, με διακυβέρνηση αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμού, Αν μου επιτρέπετε κύριε Μασούρα, έχω να σα κάνω δύο ερωτήσει για τις συστάσεις που έχετε στο τέλος τη μελέτη σα. Πρώτον, ποιο ρόλο μπορεί συγκεκριμένα να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εγκαθίδρυση ενός διαλόγου και πραγματική διαμεσολάβηση μεταξύ των κεντρικών αρχών και των περιφερειακών αρχών στο ε, Ιρακινό Κουρδιστάν. Και από την άλλη, τι πιστεύετε για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση των δυνάμεων των σωματών ασφαλείας αστυνομίας για να εσωματωθούν οι παραστρατιωτικές οργανώσεις και οι πολιτοφυλακές ε, είτε στο στρατό είτε στην αστυνομία της χώρας. Merci. Ευχαριστώ κυρία Σαϊφή. Και τώρα άλλοι συνάδελφοι. Ένας ακόμα συνάδελφος από τους Πρασίνους έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Ραϊμόν. Ραϊμόν. Είμαι Αυστριακός. Ε, δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις και έρχομαι κατευθείαν σε αυτές. Το πρώτο, ε, και στην παράγραφο 4.2 λέτε Ε, για αντικρώμενες θέσεις για το πώς θα έχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ενός ισχυρού ανδρός, ισχυροί ε, θεσμοί. Δεν κάνετε συστάσεις, δεν είναι δικιά σας δουλειά να κάνετε συστάσεις ή να προχωράτε ε, και να επιλέγετε κάτι ε, από τα δύο. δικιά μου δουλειά είναι. εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που... είναι υπέρ των ισχυρών θεσμών, όχι των ισχυρών ανδρών και των παλαιών δομών. Κατά την άποψή σας, Ποια θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθούν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί επιτόπου. Και το δεύτερο αφορά το Κουρδιστάν. Η μελέτη σας δεν γράφει το θέμα των Κούρδων του Ιράκ στο γενικότερο πλαίσιο, στα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και τη Σύρια. Εσείς πιστεύετε ότι η επιρροή της εσωτερικής πολιτικής στο Ιράκ είναι τόσο ασθενής ή ανύπαρκτη και όταν συζητάμε για το κουρδικό θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη συνολικότερη εικόνα ή όχι. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Επόμενη ερώτηση, σχόλιο. Ε, τον κύριο Κόουσο ε, που είναι αντιπρόεδρος μας και κάθεται εκεί πίσω. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μανσούρ εγώ είχα πολλές ερωτήσεις να σας κάνω. Με ενδιαφέρε το θέμα των σχέσεων της κυβέρνησης Βαγδάτης και της ε, κυβέρνησης της Κουρδικής στο Ιράκ. Μετά το δημοψήφισμα υπέρ της ανεξαρτησίας, τι απέγινε. Επίσης θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερα πράγματα για την ε, ε, ανάσταση του Άισις στο Κυρκούκ που αναφέρατε. Και η σημερινή κυβέρνηση έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα ή προσπάθησε να μην εξαιρέσει την περιοχή του Αλαμπάρ ε, από τον προϋπολογισμό. Θυμάμαι το 2011, το 2010 τον αποκλεισμό τους, που ε, αυτό οδήγησε στο να γεννηθεί το Ισλαμικό κράτος. Και επίσης ποιες είναι οι σχέσεις με την Τουρκία και το Ιράν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Άλλος. Κανείς. Όχι. Τρεις ομιλητές, πολλές ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα αρχίσω από την κυρία Σαϊφή. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε κάτι που αναφέρω στη μελέτη για τα σφάλματα που έχουν γίνει. Οι σχέσεις Ερμπίλ και Βαγδάτης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Έχουν ανοίξει και τα αεροδρόμια πρόσφατα. Έχει ληφθεί η απόφαση τουλάχιστον να ανοίξουν. Το δημοψήφισμα αυτή τη στιγμή περισσότεροι το θεωρούν ε, σφάλμα και οι ενεχόμενοι. Σας μίλησα για την ρεαλιστική ε, άποψη ενό ρεαλιστικού εθνικιστικού κινήματος σε σχέση με το ακραίο. Πολλές φορές ήταν, ε, για πολύ καιρό ήταν πολύ ρεαλιστές οι Κούρδοι. Το 2005 όταν ε, στην όταν το κράτος ε, ε, ε, οι ηγέτες ήθελαν να στείλουν τους ισχυρούς τους άνδρες στο κεντρικό κράτος. Βάλαν τον Ταλαμπανή πρόεδρο της χώρας, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έναν άλλον ισχυρό, γιατί ήθελαν να επηρεάσουν τη δημιουργία θεσμών από το εσωτερικό, του κεντρικού κράτους. Μετά το 2014 αλλά και προηγουμένως άρχισαν να αποσύρονται και αποφάσισαν ότι δεν χρειάζονται τη Βαγδάτη για να προχωρήσουν. Τι συμβαίνει τώρα στο Κουρδιστάν. Έχουν ε, συνειδητοποίησε ότι είμαστε εδώ τώρα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ε, Βαγδάτη. Και το PUK και το KDP, τα κόμματα αυτά, το έχουν καταλάβει τα κουρδικά. Από τη σκοπιά του Πρωθυπουργού του Ιράκ ε, χρειάζεται να εξετάσει διάφορα ενδεχόμενα. Αν δώσει τους μισθούς στους Κούρδους ε, στη Σουλεϊμανία και στο Ερμπίλ. Τι θα γίνει με εκείνους που είναι στη Βασόρα και είναι Σιήτες και υποφέρουν. Τι θα γίνει με τους Σουνίτες. Δηλαδή, σε κάποιο βαθμό ε, θέλησε να τους τιμωρήσει για το δημοψήφισμα, θέλησε να ενισχύσει τη δική του αξιοπιστία γιατί είναι και εκλογική χρονιά, αλλά είναι δύσκολο να δώσει τα χρήματα για όλο το Ιράκ ή σε όλο το Ιράκ ή να έρθει ταυτόχρονα οικοδόμηση και θα πρέπει να επιλέξει που θα εστιάσει. Και αυτή θα πρέπει να είναι η ευθύνη των ηγετών των Κούρδων να επιστρέψουν στην υφαλαιότητα και το ρεαλισμό που επέδειξαν στο παρελθόν. Ε, ο χρυσός αιώνας, η χρυσή εποχή των Κούρδων που μπορούσαν ε, να εξάγουν μόνοι τους το πετρέλαιο, να έχουν δικό τους αεροδρόμιο, να δίνουν βίζες, πάνε αυτά, τελειώσανε, τουλάχιστον προσωρινά. Ε, και θα πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις με το, την κεντρική ηγεσία. Ε, έχουν μάθει από τις αποτυχίες του παρελθόντος και ε, το δημοψήφισμα. Αυτό συνδέεται και με το Ιράν, διότι αμέσως μετά το δημοψήφισμα κατεβλήθη μια προσπάθεια να στραφούν κατά του Ιράν ότι το Ιράν ήταν ο κακό και οι Σιητικέ πολιτοφυλακέ ήταν ο κακό και μετά διαπίστωσαν ότι δεν γίνεται. Πρέπει να συνεργαστούμε με το Ιράν και έχει επανέλθει μια προσέγγιση. Και είναι ε, ένας ισχυρός της περιοχής ε, γείτονά σου και αν είσαι κατά του Ιράν είσαι με τους χαμένους. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο Ιράκ. Αυτό αφορά και το κουρδικό. Σε ό,τι αφορά τα σώματα ασφαλείας και ε, αυτά τα παρα στρατιωτικά, ε, παρακρατικά είναι πρόβλημα. Ε, συζήτησα με κάποιους ηγέτες του Χατζη Σάμπιτ και είπαν ότι θα πάνε αυτά τα τάγματα εκεί, αυτές οι μονάδες και τα λοιπά. Μετά τον Νοέμβριο του 2016 τώρα θεωρούν τον εαυτό τους ανεξάρτητο σώμα ασφαλείας, ένοπλο, ε, παρά τον Πρωθυπουργό. Αυτό το λέει η νομοθεσία. Και σύμφωνα λοιπόν με το Σύνταγμα αυτοί θα πρέπει να ενταχθούν ε, στο Υπουργείο Αμήνης στο Υπουργείο Ιστορικών. Τώρα είναι στον Πρωθυπουργό, με διανόμου. Και όταν το συζήτησα με την ίδια την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, είναι προηγούμενο γιατί και αυτή είναι παρά τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή και αυτή είναι σε μια γκρίζα ζώνη, παρόλο που ήταν οι πιο ε, οι, ε, οι χρυσές μεραρχίες της λέγανε στην καταπολέμηση ε, της τρομοκρατίας. Και τώρα έρχεται ε, και το CTS και λέει μπορούμε να είμαστε και μέσα για αυτούς. Χρειάζεται αναρρύθμιση. Δεν πρόκειται να ενταχθούν ούτε στο Υπουργείο Μήνης ούτε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πώς μπορεί κανείς σταδιακά να ξεφύγει από την ανάγκη να υπάρχουν αυτές οι ένοπλες ομάδες. Συναντήθηκα με έναν ηγέτη τους περισμένες εβδομάδες και μου είπε ότι η Χασίτ ήταν ε, πιο αντιπροσωπευτική γιατί έχουμε Τουρκομάνους, Γεζιδί, Χριστιανούς, είμαστε οι πιο ε, αντιπροσωπευτικοί. Θέλουν να γίνουν εθνοφρουρά ή εθνοφυλακοί, να ελέγχουν τα σύνορα κτλ. Όχι να διαλυθούν ή να ενταχθούν κάπου. Αυτές είναι οι πραγματικότητες, αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και αντί να τις και να τις παραβλέπουμε. Έτσι θα έρθει η αλλαγή. Θα στηθεί το κράτος και οι θεσμοί. Τώρα, για το άλλο που ρωτήσατε, για τους ισχυρούς άνδρες απέναντι σε ισχυρούς θεσμούς. Βεβαίως, ο καθένας ε, ήλπιζε ε, να υπάρχουν ισχυροί θεσμοί. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη να επανέλθει κάποιο τύπου Σαντάμ. Όχι, δεν θέλουν τον ίδιο το Σαντάμ, αλλά θέλουν τον θεσμό του Προέδρου. Ε, αυτό που θα πρέπει να κάνετε, όχι να στηρίξετε θεσμο, ε, προσωπικότητες, ε, ανθρώπους, πρόσωπα, αλλά τους θεσμούς και ποιον εκπροσωπούν οι θεσμοί ή ποιος εκπροσωπεί τους θεσμούς. Τώρα υπάρχει μια διάχυση εξουσίας, εντάξει υπάρχει ο Πρωθυπουργό ε, που ενδιαφέρεται πολύ για αυτό το, το τομέα. Αλλά ε, ολόκληρη δομή εκεί υπάρχουν κρατικές δομές, ημικρατικέ, παρακρατικές, υβριδικέ και όλοι έχουν εξουσία. Θα πρέπει να οικοδομηθούν θεσμοί και να ξεφύγουμε ε, από πρόσωπα. Να μιλάμε το Υπουργείο του ΤΑΔΕ ή η Επιτροπή του ΔΗΝΑ. Το κουρδικό τώρα και το ευρύτερο. Πολλοί ηγέτες του κουρδικού, ιδιαίτερα από το κόμμα και είχαν πολύ καλέ σχέσει με την τουρκική κυβέρνηση. Οικονομικές σχέσεις και εμπόριο κάνανε. Δηλαδή, και τώρα έχουν μεγάλο πρόβλημα με το ΠΚΚ και το PYD. Αυτή η ιδέα του μεγάλου Κουρδιστάν σε κάποιο βαθμό ε, έχει προβληθεί υπερβολικά. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα που έχουν μεταξύ τους τα κουρδικά κόμματα με τη Συρία, με την Τουρκία και με το Ιράκ. Και το ΠΚΚ ε, δραστηριοποιείται και ε, στην Ινεβή και στο Σιντζάρ και σε άλλα μέλη του Ιράκ. Παίζει το ΠΚΚ ρόλο. Για τον Τάες, το ISIS, το Κυρκούκ. Το Ισλαμικό κράτος ως οργάνωση ξεκίνησε στο Αμπάρ. Από εκεί άρχισαν ε, ε, να δίκουν και μετά πήγαν στη Μουσούλη και μετά ε, τους διώξαν από εκεί και ψάχνουν νέα εδάφη. Πού θα βρουν αυτά τα νέα εδάφη εκεί που υπάρχουν συγκρούσεις, εκεί που υπάρχει κενό εξουσίας. Κυρκούκ και γύρω-γύρω υπάρχουν ε, κέντρα τεράστια οικονομικά. Το υπαριθμόν ένα κίνητρο είναι οικονομικό περισσότερο από η ιδεολογία, οικονομικό και εξουσία. Εκεί λοιπόν που έχετε ομάδες αντικρώμενες, έχετε τους ΠΕΣΜΕΡΓΑ, την αστυνομία, ομοσπονδιακή, τοπική, παραστρατιωτικές οργανώσεις, χάος επικρατεί εκεί. Ε, κάθε μέρα βγαίνουν, φυτρών νέα φυλάκια που κάνουν ελέγχους. Ε, δεν ξέρει κανείς που πηγαίνει η περιοχή. Έχει αποσυρθεί το κράτος από την περιφέρεια αυτή και είναι πρόσφορο έδαφος για να αναδυθούν ομάδες τύπου ISIS. Δηλαδή μπορεί κάπου να ιτηθείς, να φύγεις από μια πόλη, αλλά να ξεφυτρώσεις κάπου αλλού. Και ο ρόλος του Ιράν και της Τουρκίας, όπως σας είπα το Ιράν, έχει βαθιές ρίζες στο Ιρακινό κράτος στην Ουάσιγκτον ίσως υπερβάλλουν ως προς το ρόλο του ε, Ιράν. Το Ιράν όμως δεν θέλει το Ιράκ να διαλυθεί, θέλει να είναι εταίρος, μικρότερος, ωστόσο εταίρος. Από το 2014 έμαθαν ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τις σκεφτικές πολιτικές ε, αυτές καθ' αυτές, γιατί ε, θα έρθει και άλλο ISIS που δεν θέλει ο Ιράν αλλά το Ιράν ε, ελέγχει πολλούς ε, ηθήνοντες ή μη κρατικούς ε, ομάδες ένοπλες κτλ. Αλλά το Ιράν δεν είναι κοντόφθαλμο, έχει μακρά προοπτική. Παράδειγμα, στο δημοψήφισμα στο Κυρκούκ, όταν λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκέ χώρε ήταν πεπισμένοι ότι ο πρόεδρο Μπαρζάνικα με κάποιο τρόπο θα το ανέβαλε το δημοψήφισμα ή θα το ματέωνε δεν κάνανε κανένα σχέδιο συγκράτησης και, και αντιμετώπισης τι θα γίνει αν θα γίνει το δημοψήφισμα. Το Ιράν το κατάλαβε πολύ περισσότερο και είχε σχέδιο καταστρώσει πριν το δημοψήφισμα γιατί ήξερε ότι θα γίνει το δημοψήφισμα. Και πέρσι τον Οκτώβριο όταν προσπαθούσαν οι ΗΠΑ να καταστρώσουν κάποια σχέδια το Ιράν είχε δικό του, γιατί έχει μακρά ε, προοπτική, μακρινή ματιά. Η Τουρκία προσπαθεί τώρα να δυθεί, έχει πολλή δουλειά στη Συρία και εσωτερικά, αλλά στην Ινωβή και στην, ε, στην Ευή, συγγνώμη, και στη Μοσούλη και στο Κυρκούκ προσπαθεί να διατηρήσει την επιρροή της, γιατί είναι στα σύνορά της. Ευχαριστούμε κύριε Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, σχόλια. Όχι. Ωραία, ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε εδώ. Ε, ε μένετε στο Λονδίνο, ε, δεν κάνω λάθος. Ναι, ωραία λοιπόν, καλό σας ταξίδι, καλή επιστροφή. Διακόπτουμε τώρα και θα συνεχίσουμε στις 2.30. Και ελπίζω ότι ο αντιπρόεδρος μας, ο κ. Κόσο, θα μπορέσει να προεδρεύσει την συνεδρίαση. Καλή σας όρεξη.